Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι και καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας. Η τελευταία μας ε, πριν από τις καλοκαίρινες διακοπές και αύριο βέβαια θα συνεδριάσουμε. Ε, είμαστε πολύ εδώ σήμερα γιατί έχουμε και ψηφοφορία. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Δεν ε, βλέπω να ζητάει κανείς αλλαγή. Συμφωνείτε, εγκρίνετε. Καλώς. Και περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης, εκλογή δεύτερου ή δεύτερης αντιπροέδρου. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, ο Πάβο Βάιρινεν, που ήταν ο αντιπρόεδρός μας, πάει στο Φιλανδέζικο Κοινοβούλιο τώρα και πρέπει να τον ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για το έργο του εδώ στην Επιτροπή μας. Ασχολήθηκε με πολλές εκθέσεις, με θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά. Συνεπώς, ποιος μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος. Ε, υπάρχουν ονόματα για αντικατάσταση. Προτείνει τον κύριο Πόγκα ο κύριος Βίλαντ. Αντικαθιστά τον κύριο Βέντα. Και ο κύριος Ρούμπεκ, τον κύριο Πρέντα, όσον αφορά την ψηφοφορία. Έτσι από το άλλο. Οι σοσιαλιστές. Ο Ρίκε Κερέρο. Αντικαθίσταται από τον Χωσέ Μπλάνκο. Και ο Βίνσεντ Πεγιό από τον κύριο Μασκούρ. οπότε υπάρχουν διάφοροι αναπληρωτές. Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα έπρεπε να ξέρω ότι αντικαθιστά. Βλέπω ότι έχουμε απαρτία, χρειαζόμαστε το 1 τέταρτο των μελών για να είναι έγκυρη η ψηφοφορία. Συνεπώς, υποψήφι τώρα για τη θέση της πρώτης, της δεύτερης, συγγνώμη, διορθώνει πρόεδρος, αντιπροεδρίας της δεύτερης αντιπροεδρίας, γιατί έχουμε εδώ τον πρώτο αντιπρόεδρο. Λοιπόν, υποψήφι για τη θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου, παρακαλώ. Παρακαλώ. Η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ναι, με ιδιαίτερη χαρά. Προτείνω την Μύρια Δέκα Πέρα στην ε, θέση του δεύτερου αντιπρόεδρου. Γνωρίζω τη συνάδελφο εδώ και πολλά χρόνια από τη συνεργασία που είχαμε και στο Φιλανδικό Κοινοβούλιο. Ωραία, υπάρχει η υποψηφιότητα αυτή της κυρίας Βέκα Πέρα. Παρακαλώ, και εσείς έχετε κάτι να πείτε, κύριε Γκέρενς. Ναι, και εγώ προτείνω τη συνάδελφο γιατί είναι από την ομάδα μου. Απλώς άφησα προτεραιότητα στις γυναίκες, έτσι πρώτα να το προτείνει μια γυναίκα, αλλά την προτείνω κι εγώ. Καλώς άλλες πολιτικές ομάδες, οι 5% των μελών έχουν να προτείνουν άλλον υποψήφιο. Όχι από ό,τι βλέπω. Οπότε η κυρία Βέκα Πέρα συμφωνεί να είναι υποψήφια. Καλώς. Ωραία. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Αλλά πρώτα πρέπει να διαβάσω κάτι άλλο. Περιμένετε γιατί πρέπει να κρατήσουμε τους τύπους, έτσι πρέπει να επενθυμίσω στην υποψήφια ότι πρέπει να είναι πλήρες μέλος της Επιτροπής αυτής που είναι και ότι πρέπει να έχει συμπληρώσει και τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων της. Το έχετε κάνει? Ωραία. Αφού δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος λοιπόν, ε, προτείνω την εκλογή διαβοής της ε, συναδέρφου Φεκαπέρα. Θέλετε μήπως να πείτε κάτι, θέλετε κάτι να πείτε, να συστηθείτε, να μας παρουσιάσετε τον εαυτό σας. Ευχαριστώ πολύ. Να ξέρετε ότι με χαρά είμαι μέλος της Επιτροπής αυτής Ανάπτυξης και δεύτερη αντιπρόεδρος. Και όπως είπατε ήδη, ο κύριος Πάβο Βάιρινερ πήγε στη Φιλανδική Βουλή. Οπότε ουσιαστικά αλλάξαμε θέσεις. Εγώ ήμουνα 11 χρόνια στο Φιλανδικό Κοινοβούλιο και τώρα είμαι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα θα έχουμε πολλά να κάνουμε σε σχέση με τη μετανάστευση, το προσφυγικό, τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ένα τεράστιο θέμα αυτή τη στιγμή. Μας μένει ένας χρόνος. Οπότε εγώ είμαι γεμάτη ενέργεια να δουλέψω στην Επιτροπή αυτή και προσβλέπω στην ε, καλή συζήτηση και καλή συνεργασία που θα έχουμε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω επίσης στη θέση της δεύτερης αντιπρόεδρου. Μπορείτε να έρθετε εδώ, να καθίσετε στο βήμα. Οπότε αλλάξτε θέση, εδώ είναι η θέση σας. Λοιπόν, πάλι χειροκρότημα για τη συνάδελφο. Ωραία, σημείο 3. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Δεν έχω ανακοινώσει. Σωστά. Και περνάμε στο σημείο 4. Έγκριση των αποφάσεων και των συστάσεων των συντονιστών. Οι αποφάσεις και οι συστάσεις είναι στους φακέλους σας. Ε, έχετε τίποτα να σχολιάσετε, αν ναι, στη γραμματεία παρακαλώ πριν τη λήξη της συνεδρίας αυτής. Τώρα, Επιτροπή έχει ανακοινώσει όχι, δεν ε, ξέρω τίποτα τέτοιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχουμε καμία ανακοίνωση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και συνεπώς συνεχίζουμε και περνάμε στην ψηφοφορία. Σημείο 6 στην ημερήσια διάταξη, μία ψηφοφορία έχουμε, αυτή μόνο, που είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεσμευτικό χαρακτήρα μέσω του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις με διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνήσαμε να συντάξουμε ψήφισμα πριν τον Οκτώβριο, τη συνάντηση του ΟΗΕ δηλαδή του Οκτωβρίου. Η βασική ιδέα είναι ότι θα ψηφίσουμε τώρα εδώ και το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Και θα έχουμε και κοινή συζήτηση με την ΙΝΤΕ και την Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για προφορική ερώτηση προς την ε, Αντιπρόεδρο και Υπατικπρόσωπο. πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους για τη συμβολή τους στο φάκελο αυτό. Και περνάμε ευθύ αμέσω στην ψηφοφορία. Μπορεί να κρατήσει πολύ, θα δούμε, εξαρτάται, εξαρτάται. Έτοιμοι, αρχίζουμε λοιπόν. Συμβαστική 13, πρώτα απ' όλα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε για την 114. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 114 λέει πάλι πρόεδρος. Α, συγγνώμη, διορθώνει. 115 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σας υπενθυμίζω συνάδελφοι, ότι μερικές ψηφοφορίες όπως 116 και κάποιες άλλες έχουν δίπλα ένα και γραφημένο είναι γιατί έχουν αλλάξει κανόνες και επειδή οι συνάδελφοι αυτοί δεν είναι μέλη της Επιτροπής μας δεν μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες εξού και δεν θα τις ψηφίσουμε. 117 λοιπόν η επόμενη ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ υπέρ κατά αποχές. Ποιος, ε, για το ΕΛΚ ποιος ε, δίνει την κατεύθυνση. Λοιπόν, 115, συγγνώμη, συμβαστική 15, ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Με μεγάλη διαφορά. Να ξέρω ποιος δίνει την κατεύθυνση από το ΕΛΚ. Εκτός μικροφώνου η παρέμβαση του κύριου Έγγελ. Τελευταίο τμήμα της 123 ε, παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές δεν βλέπω πώς ψηφίζουν οι μάτες θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν παρακαλώ ψηφίστε 18 συμβαστική 18 ψηφίστε παρακαλώ πέρας εγκρίθηκε με μεγάλη διαφορά Συμβαβεστήκε 19 επέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. Η ηλεκτρονικά. 146. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Α, από το ΕΛΚ ψηφίζουν ένας παραπάνω. Λοιπόν, για σταματάμε την ψηφοφορία εδώ. Μια στιγμή. Πρέπει να διορθωθεί αυτό. Έχουμε έναν παραπάνω από το ΕΛΚ. Λοιπόν, 8 Πρέπει να είναι από το ΕΛΚ. Έβγαλε ένα στην κάρτα του. Έτσι είναι οι κανόνες. Λοιπόν, ξαναψηφίζουμε. Πού ήμασταν? Τροπολογία 146 του Λί Μισελ. Υπέρ παρακαλώ. Λέει πρόεδρος, αλλά διορθώνει, όχι, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 146. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ. Ποιος από το ΕΛΚ. Ποιος από το ΕΛΚ δίνει την κατεύθυνση. Για να βλέπω, να ξέρω. Αλλιώς αργούμε πολύ. Πρέπει να ξέρω τι κάνετε. «148 απορρίφθηκε. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, νομίζω και απορρίπτεται, λέει Πρόεδρος. Μπορείτε να ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίφθηκε. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 158, ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Και απορρίπτεται. Εκατόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 160 και 161 μαζί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 162, όχι καταπίπτει. 163 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 165 υπέρ, ...165 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 177 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε για την 179. Ωραία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 179. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Ισοψηφία. Κα... Άρα απορρίπτεται. Εντάξει, δίκιο είχατε. Απορρίφθηκε. Ναι, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. 168 υπέρ. Υπέρ κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά 168. Ψηφίστε. Πέρας. Απορρίφθηκε. 181 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, νομίζω ότι απορρίπτεται. Αλλά ε, ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίφθηκε. 185 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 186 απορρίφθηκε, ε, συγγνώμη, έχει αποσυρθεί. 2 επιστηματική υπέρ, κατά, 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 50. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της προφορίας απορρίφθηκε. Έκανα λάθος, λέει ο κύριος Ντέβα. Δεν γίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 52. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 53 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 53 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Είναι δύσκολο να δω. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να δείχνουν οι ομάδες τι λένε. Λοιπόν, συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές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 απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 81. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραση της η Ισοψηφία απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά και για την 82. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. The Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 93 υπέρ. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία όχι, ναι, τροπολογία 100 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε ηλεκτρονικά έναρξη της ψηφοφορίας. Ψηφίζατε όλοι, Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. εποχέ. απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Μπορεί το ΕΛΚ να δείξει τι ψηφίζει. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. αποχέ. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Ας κλείσουμε την προηγούμενη συμφορία. Ωραία. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαληθεύουμε την 9. Λήξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά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 31 υπέρ. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του ψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. 15 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλες ψηφοφορίες. Προχωράμε. Προχωράμε. Γιατί έχουμε, έχει σειρά προπολογισμό. Παρακαλώ πολύ, αν θέλετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα ήσυχα. Σημείο 7 τη ημερήσια διάταξη. Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτο 2019. παρακαλώ πολύ, αν θέλετε να συζητήσετε εκτός της αιθούσης. Ευχαριστούμε, Τερέζα. Okay, colleagues, we're, um, we're going to move on to... Περνάμε στην γνωμοδότηση για τον προπολογισμό. Τον Απρίλιο ήδη ανταλλάξαμε απόψη με τον Ντανιέλε Βιώτη, τον εισηγητή της Επιτροπής Προπολογισμών. Αυτό που συζητάμε ε, συμπεριλαμβάνει και το ο, χρηματοδοτικό όργανο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Η εισηγήτριά μας είναι η Άρνε Λίτς, ε, η οποία έχει προτάσεις σε σχέση με, την, με το κείμενο που έχει υποβάλει ο κύριος Βιώτη. Ο, ο, συγγνώμη, ο Αρνελίτ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Να πω πως ε, χθες έγινε και μία ακρόαση μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους ναι. στόχους ε, βιώσιμης ανάπτυξης και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα κρόσα γιατί είδαμε όλα αυτά που γίνονται πάνω στο θέμα αυτό. Προσπάθησα λοιπόν ε, στη γνωμοδότηση για τον προπολογισμό να ε, τονίσω το ρόλο της εκπαίδευσης, της υγείας, της ισότητας των φύλων και της κλιματικής δράσης. Αυτά είναι τα σημεία επιγραμματικά και θα ξεκινήσω λοιπόν με την παρουσίαση της γνωμοδότησης λέγοντας ότι είναι η ανθρωπιστική βοήθεια βασική. Τα κράτη-μέλη πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για να αυξήσουν την αναπτυξιακή βοήθεια στο 0,7 του καθάριστου εθνικού εισοδήματος μέχρι το 2030. Χρειάζεται λοιπόν να αναφερθεί το θέμα αυτό, αλλά και να υπάρχει εξαίρεση του κόστου ε, των ε, δωρητών ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε εκ νέου το θέμα του χρέους. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τους ε, εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους πρέπει επίσης να εξεταστεί και να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό Επίσης, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να χρηματοδοτεί και την εκπαίδευση και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή, αν μπορεί να μου απαντήσει, εάν υπάρχουν τα στοιχεία αυτά για την ε, χρηματοδότηση της εκπαίδευσης ε, μέσω της ανθρωπιστικής βοήθειας και πού βρισκόμαστε, να μας πει μερικά ε, στοιχεία. Έχουμε μεγάλη και μακρά ιστορία ανθρωπιστικής βοήθειας. Είναι πάνω από 20 ετών τα προγράμματα και πρέπει λοιπόν να επανασχεδιαστούν. Τα κονδύλια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως για παράδειγμα ελέγχου στα σύνορα. Αυτό έχει τονιστεί και ε, στο πλαίσιο της συζήτησης τη χρήση των πόρων του καταπιστεύματος για την ε, Αφρική. Χρειάζεται επίση να ενισχυθεί η κλιματική διπλωματία και η γνώση και η μεταφορά αυτής Επίσης, συνομίλησα με εκπροσώπους της Γενικής Διευθύνσης ΝΙΑΡ και έμαθα ότι η ανθρωπιστική βοήθεια, το νερό για την ακρίβεια δεν χρησιμοποιείται στο 100% αλλά υπάρχουν μεγάλες διαρροές. Είναι πολύ Σημαντικό λοιπόν να ενισχυθεί η κλιματική διπλωματία και η χρηματοδότηση έργων για ε, το κλίμα στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης, ε, αναφέρεται η ανάγκη αναθεώρησης του κανονισμού για την ανθρωπιστική βοήθεια, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κλιματική διπλωματία. Επίσης, αναφέρεται η κατάσταση στην και στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά παραθέτω την ε, παράγραφο αυτούσια που τονίζει ε, την ε, ανάγκη ενίσχυσης της Ούνρα και της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Ούνρα πρέπει λοιπόν να στηριχθεί για το συμφέρον όλης της περιοχής. Αυτό το έχει τονίσει και ο στρατός του Ισραήλ. Τώρα, σε, ε, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει ιδιαίτερε περικοπές, όμως εμείς ε, ζητούμε την προσθήκη επιπλέον πόρων για ανθρωπιστική βοήθεια, μια που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυτή η αύξηση του 15%. Ε, που διοχετεύεται κυρίως στις εγκαταστάσεις για τους πρόσφυγες στην Τουρκία, όμως αναφέρεται και το θέμα των υπόλοιπων χωρών. Τι γίνεται στη Συρία, τι γίνεται στο Λίβανο, όπου παρατηρούνται εντάσεις και εντός ε, το, της ε, χώρας. Ζητούμε επίση υψηλότερο αποθεματικό έκτακτη βοήθεια, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο γρήγορα σε κρίσει. και ζητούμε το ίδιο επίπεδο πιστώσεων πληρωμών με την πιστώσει υποχρεώσεων έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά στη χρηματοδότηση. Εδώ να ευχαριστώ τους συναδέλφους Γκερέρο και Τελειών και τους ε, βοηθούς ε, αλλά και τον Σάρλ Γκέρντς για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Αναφέρω στην εκνομοδότησή μου και τη θέση του Συμβουλίου που έχει προτείνει περικοπές ε, πληρωμές και υποχρεώσεις των DCI ε, και ζητούμε λοιπόν αναθεώρηση. 18 Ιουλίου είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών και λόγω των θερινών διακοπών θα περιμένουμε τις απαντήσεις των ε, συναδέλφων μετά. Ελπίζω λοιπόν η γνωμοδότησή μας να οδηγήσει σε μια ε, ισχυρή θέση της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Περάσουμε, θα περάσουμε τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Ρούμπιγκ έχει το λόγο εκ μέρους του ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω λοιπόν και εγώ τον συνάδελφο Αρνελίτς, διότι νομίζω πως έχει αναφέρει όλα τα σημαντικά ε, στοιχεία και τις θέσεις της Επιτροπής μας για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η στόχη αυτή είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις της αναπτυξιακής πολιτικής, της χορήγησης ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Η υγεία λοιπόν, η εκπαίδευση, η κλιματική στόχη είναι πάρα πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα στο τομέα της εκπαίδευσης η, η εκπαίδευση για την ισότητα των φύλων είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό είναι από εξίσου σημαντικό στη δεύτερη φάση των ε, στόχων των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης να τονιστεί η διάσταση της ισότητας. Νομίζω πως ε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε παρατηρώντας την κατάσταση πως ε, υπάρχουν προβλήματα που πρέπει, μπορούμε για παράδειγμα να στηρίξουμε τις προσπάθειες που γίνονται τόσο για την ε, γεωργία και την άδευση όσο και για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα μας παρέχει τις λύσεις, έχει τεράστιο δυναμικό και ε, επίσης η βελτίωση των υγειονομικών συνθήκων, ε, της ίδρευσης θα είναι πάρα πολύ σημαντικές. Στα νοσοκομεία υπάρχει πρόβλημα. Το 50% των νοσοκομείων έχουν ε, μολυσμένο νερό. Αυτό σίγουρα δεν είναι καλό και πρέπει να αλλάξει. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό να δούμε αυτή τη διάσταση αλλά και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Όλοι οι στόχοι αυτοί έχουν αναφερθεί και στις προηγούμενες συνόδους για την αναπτυξιακή βοήθεια και νομίζω πως ε, ταιριάζουν μεταξύ τους και είναι πολύ σωστό που αναφέρονται στη γνωμοδότηση. Θα μας απασχολήσουν εξάλλου και στο μέλλον. Δεύτερον, αυτό που μάθαμε με τα Ταμεία Συνοχή στην Ευρώπη είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να στοχεύουμε στις επιμέρους περιφέρειες σε μικρά έργα, να χρηματοδοτούμε και να στηρίζουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έτσι ώστε να υπάρχουν συνέργειες, να χρηματοδοτούμε επίσης και να στηρίζουμε την επαγγελματική κατάρτιση, την επανακατάρτιση, έτσι ώστε αυτό, αυτή η στήριξη έργων σε τρία στάδια, τον εντοπισμό δηλαδή, τη στήριξη και την ε, μετεκπαίδευση, να βοηθήσει σε στη βελτίωση των ε, συνθήκων στο μέλλον. Επίσης, οι δημόσιοι διαγωνισμοί πρέπει να ε, γίνουν ε, με βελτιωμένο τρόπο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των επενδύσεων για τους πολίτες. Στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού έχουμε δει περιπτώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πάμε σε μια περιφέρεια χρηματοδοτείται ένα έργο, μια εγκατάσταση, όλα είναι πολύ καλά μέχρι να δούμε στην ουσία τι συμβαίνει, τα προβλήματα που υπάρχουν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να δούμε τα θέματα αυτά όπου χρήζουν βελτίωσης. Ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, μπορούμε να κάνουμε πολλά και να τις στηρίξουμε. Να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε τόσο καλά και αυτήν την έκθεση ε, του προπολογισμού. Εμείς φυσικά θα στηρίξουμε τις ε, προτάσεις σας στο μέτρο του δυνατού. Αλλά να πούμε και ότι δεν γίνεται τίποτα χωρίς διεθνή συνεργασία. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες από όλες τις πλευρές. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Αρνηλίτση για την γνωμοδότησή του η οποία αναφέρει όλα αυτά τα πολύ σημαντικά σημεία. Η κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κατά. Ε, καταρχήν θα ήθελα να, ε, να διαχωρίσουμε ξεκάθαρα την ανθρωπιστική από την αναπτυξιακή βοήθεια. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να τα σμίγουμε. Η ανθρωπιστική βοήθεια παρέχεται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και όταν υπάρχει εξαιρετικά επίγον λόγος. Βεβαίως η εκπαίδευση είναι το α και το ω της ανάπτυξης και αυτή θα πρέπει να είναι στην ε, πρώτη γραμμή δεδομένου ότι βοηθούμε τους ανθρώπους να επιβιώσουν γιατί ένας νεκρός δεν μπορεί να εκπαιδευτεί. Ε, τώρα, όσον αφορά την χρήση ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση υπάρχουν πολλοί ε, πολλές ευκαιρίες για να χρησιμοποιηθεί, όπως για παράδειγμα τα εκτοπισμένα παιδιά. Ήμασταν με την κυρία Πρόεδρο στην Ουγκάντα και είδαμε ότι τα παιδιά των εκτοπισμένων από τον Νότιο Σουδά δεν είχαν τη δυνατότητα εκπαίδευσης. Εκεί όντως η ανθρωπιστική βοήθεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση τους. Επίσης, σε διάφορα μέρη, σε πάρα πολλά μέρη της Αφρικής, τα σχολεία δεν λειτουργούν λόγω υποσυτισμού των ε, παιδιών, λόγω έλλειψης σχολικών ειδών. Πολλά παιδιά δεν έχουν ούτε ένα μολύβι και το πιο ωραίο δώρο που μπορείς να τους κάνεις είναι ένα μολύβι, ένα τετράδιο. Ε, πάνε ξυπόλυτα στα σχολεία. Νομίζω ότι σε αυτό το τομέα θα πρέπει να προσδιορίσουμε τη δυνατότητα να βοηθηθούν τα παιδιά. Θέλω να κάνω και το ζήτημα των εμβολιασμών φυσικά οι οποίοι ναι μεν παρέχονται δωρεάν για τα μικρά παιδιά αλλά δεν υπάρχει ο μηχανισμός εκείνος που θα, ε, θα βοηθήσει τα παιδιά να δεχθούν τους εμβολιασμούς. Θέλω να επισημάνω ένα γεγονός ότι λόγω της διαφθοράς και της άκρα της γραφειοκρατίας που υπάρχει στην Αφρική σε πολλές περιοχές όπου έχουμε ιδρύσει σχολεία με ε, private donors, με ιδιωτικές δωρεές, μας υποχρεώνουν για κάθε δύο παιδιά να κατασκευάζουμε και μία τουαλέτα. Ενώ εγώ δεν γνωρίζω σχολείο της Ευρώπης που να υπάρχουν περισσότερες από μία τουαλέτα ανά 50 παιδιά, ανά 40 παιδιά. Αυτή είναι η αναλογία. Προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα, μπας περιπτώσει, να κλέψουν περισσότερα χρήματα. Δεν διστάζω να πω αυτή τη φράση γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτό τον τομέα ίσως θα έπρεπε να είχαμε μια ισχυρότερη παρέμβαση. Δηλαδή για να λειτουργήσει ένα σχολείο με 2.000 μαθητές μας υποχρεώνουν να κατασκευάσουμε 800 τουαλέτες. Ε, Άλλο πάρα πολύ σημαντικό το οποίο μπορεί να ενταχθεί και στα πλαίσια του 0,7% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος το οποίο πρέπει να δίνεται για αναπτυξιακή βοήθεια. Σε αυτό ειδικά για τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης οι οποίες όμως έχουν και ένα υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο θα μπορούσε να ενταχθεί η δυνατότητα εκπαίδευσης παιδιών από υποανάπτυκτες χώρες, μάλλον ε, φοιτητών είτε ε, γιατρών για παράδειγμα για την ε, απόκτηση εξειδίκευσης ε, προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα τους και να είναι χρήσιμοι στην περιοχή από την οποία κατάγονται. Αυτό ουσιαστικά δεν κοστίζει τίποτε στην Ευρώπη. Και dormitories υπάρχουν μέσα στα νοσοκομεία και ένας επιπλέον ειδικευόμενος δεν θα παρενοχλήσει το όλο σύστημα εκπαίδευσης γιατρών. Αν μιλάμε για γιατρούς το ίδιο ισχύει και για τους δασκάλους που είναι ό,τι, ό,τι περισσότερο χρειάζεται η Αφρική και για τις νοσοκόμες και για τις ε, μαμές, για τις ε, midwives, για τους μεταφραστές. Εν πάση περιπτώσει ε, θα κάνω τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό που έχετε κάνει και θα τα ξαναπούμε. Yes, thank you. Just remind... Ευχαριστούμε πολύ. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε για το θέμα των μεών μια έκθεση πρωτοβουλίας και θα το συζητήσουμε αύριο. Το θέμα της εκπαίδευσης σε έκτακτες καταστάσεις είναι ένα ζήτημα, αλλά υπάρχει και το θέμα της εκπαίδευσης γενικά, πώς γίνεται σε μεγάλες τάξεις με πάρα πολλά παιδιά που δεν υπάρχουν μέσα, διευκολύνσεις και τελικά η δυνατότητα να εκπαιδευτούν. Ακούσαμε ένα δάσκαλο να λέει ότι τελικά με τόσα πολλά παιδιά ε, την πειθαρχία προσπαθούσε να επιβάλλει μόνο, δεν κατάφερνε να διδάξει. Οπότε δεν ξέρω. Αύριο το πρωί πρέπει να το ρωτήσουμε αυτό. Δεν ξέρω αν θα μπορούμε να έχουμε απάντηση και αν κάποιος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να μας βοηθήσει αύριο. Ας ελπίσουμε στο θέμα του κύριου Παρακαλώ, Άλντε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να στηρίξω εκ μέρους της ομάδας μου τις προτάσεις που έγιναν από τον συνάδελφο Άρνε Λίτς. Έχω τέσσερις παρατηρήσεις, επιτρέψτε μου. Η πρώτη μου έχει να κάνει με την πρώτη πρόταση που είναι στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Δηλαδή, όταν μιλάει για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης του 2030. Θα ήθελα να προσθέσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το έχει σαν στρατηγική προτεραιότητα και να αντικατοπτρίζεται αυτό στον προπολογισμό. Συμφωνώ και με το δεύτερο σημείο που μιλάει για την χρήση των αναπτυξιακών πόρων για άλλες χρήσεις πέρα από τις αναπτυξιακές και έχω και μια παρατήρηση όμως για το τρίτο σημείο ο Άρνε προτείνει να βγάλουμε από τον υπολογισμό του δημόσιου χρέου την αναπτυξιακή βοήθεια. Μένα δεν με προβληματίζει αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν αναφέρεται στο διοικητικό κόστος. Αν θέλει να κάνει διάκριση ανάμεσα στο διοικητικό κόστος και το κόστος το οποίο ε, προκαλείται στις χώρες ε, δωρητές όταν πρόκειται για τη χρηματοδότηση, δηλαδή ανταλλαγών, υποτροφιών, ε, εμπειρογνωμόνων που έρχονται από τις βονάπτυξη χώρες σε εμά. Ε, όλα αυτά είναι δαπάνες που γίνονται σε εμά βέβαια, αλλά έχουν αναπτυξιακό σκοπό. Κατά τη γνώμη μου το σημαντικό είναι η ποιότητα της προσπάθειας που μετράει. Πολύ περισσότερο από ότι το που πληρώνεται. Για την υποδοχή των προσφύγων έχω άλλη άποψη. Κάποιες χώρες το βάζουν στη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια, άλλες όχι. Θα ήταν καλό πάντως να προσθέσουμε και κάτι για μετά το Brexit. Του χρόνου είναι η πρώτη χρονιά όπου το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλήρες μέλος. Και από ό,τι έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή μας, θα έπρεπε να φροντίσουμε οι σχέσει μας με τον Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνουν όσο γίνεται πιο στενές. Αυτά. Επαναλαμβάνοντας ότι στηρίζω πλήρω το έργο του συναδέλφου Άρνε Λίτς. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ για το τρίτο που είπατε. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Γιατί θα πούνε τα μέλη τη Επιτροπή Προπολογισμών ότι αυτό έχει να κάνει με τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και όχι με τον Προπολογισμό των χωρών μελών. Λοιπόν, η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από ό,τι άκουσα από τον εισηγητή και από τις άλλες πολιτικές ομάδες, βλέπω ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα αρχίσω με κάποιες θετικές παρατηρήσεις. Βλέπω ότι η ανάλυση του φύλου θα γίνεται πλέον συστηματικά η διάσταση του φύλου, δηλαδή για όλες τις εξωτερικές δράσεις και στα διμερή και στα πολυμερή προγράμματα. Αυτό αποτελεί σίγουρα μια καλή πολιτική δέσμευση που αναλαμβάνουμε. Η ανθρωπιστική βοήθεια, καλός κακός, χρειάζεται όλο και περισσότερο. Ε, θα υπάρχουν όλο και περισσότερες ανθρωπιστικές κρίσεις και πρέπει να είμαστε σε θέση να αποκρινόμαστε. Τώρα όταν πάμε όμως στην υλοποίηση των στόχων της χιλιετίας, εκεί ε, είμαστε πιο επικριτικοί. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της ε, τώρα του στόχους του 2030, περισσότερο εξηγώντα ε, σε ποιους στόχους της χιλιετίας συνεισφέρει το κάθε πρόγραμμα. Δεν βλέπω όμως ένα πραγματικό σημάδι για αλλαγή νοοτροπίας, για αλλαγή προτύπου, πώς δηλαδή λαμβάνονται πράγματι υπόψη οι στόχοι της χιλιετίας. Και δεν νομίζω ότι, και αναπτυξιακή δεν νομίζω ότι πρέπει να το φροντίσουμε και μάλιστα ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, και όσο γίνεται πιο γρήγορα πρέπει να ξεκινήσει. Βλέπουμε επίση ότι έχουμε τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ που θα σήμαινε ότι μπορούμε να ξοδέψουμε τόσα παραπάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως μάλλον δεν έχει αυτή την πρόθεση και καλό θα ήταν να τη ρωτήσουμε γιατί. Τώρα όσον αφορά τις γραμμές στον προπολογισμό για την αναπτυξιακή βοήθεια, τα προγράμματα παραμένουν λίγο πολύ το ίδιο. Για τη Λατινική Αμερική υπάρχει μια αύξηση 3,6%. Νότια Αφρική 11,5% και Μέση Ανατολή 133% αύξηση. Καλό θα ήταν να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί. Φυσικά και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ε, νέου είδους πολύπλευρες κρίσεις στην περιοχή, αλλά 133% αύξηση ε, είναι χωρίς προηγούμενο. Η Επιτροπή λέει ότι 23 εκατομμύρια η είναι δεν ξέρω, λέει η ομιλήτρια. Μίλιον. Εκατομμύρια για το Ιράν, Ιράκ και την Ιεμένη. Αλλά τα 88 εκατομμύρια παραπάνω δεν ξέρουμε πού θα χρησιμοποιηθούν, πώς. Συνεπώς, μπορούμε να επικεντρωθούμε στο θέμα του πώς η στάση αυτή απέναντι στους ε, στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θα αλλάξει και θα συμπεριληφθούν. Και πρέπει να αναφερθεί και ο στόχος του 5%. Είναι βέβαια ένας συνδυασμός συνεισφοράς χωρών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι από το οποίο δεν πρέπει να παραιτηθούμε. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλου συναδέρφου από την Επιτροπή που μα ζητούν το λόγο. Κάποιε ερωτήσει απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ κανέναν από την Γενική Διεύθυνση ΑΦΚΟ. Έχουμε. ΔΕΦΚΟ, συγγνώμη, ανάπτυξη. Μπορεί κανεί να απαντήσει για την αύξηση αυτή σε διάφορες γεωγραφικές περιοχέ. για παράδειγμα. ποιο είναι εδώ, ο κύριος Α, προηγουμένω ή στο τέλο θα, στο θα σας δώσω το λόγο, ε, στον εισηγητή, αλλά πρώτα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ή θέλει τώρα να κάτι να προσθέσεις. Όχι, στο τέλος. Στο τέλος θα σα δώσω το λόγο, Βεβαίω. Ναι. Οπότε. Ντανιέλε Νταμίκο. Ε, σωστά, εσείς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον προπολογισμό. Ωραία. Παρακαλώ. Την τεύκο είστε, έτσι δεν είναι. Ναι. Έχουμε και την ΕΚΟ βέβαια. Ακούσαμε με πολύ προσοχή όσα έθιξε η συγγήτρια και η άλλη συνάδελφή σας. Ως γενικό σχόλιο θα έλεγα ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε να σεβαστούμε τις προτεραιότητες ε, του, των όσων έχουν σχέση με το μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής ε, συνεργασίας και τις προτεραιότητες δηλαδή τις τις οποίες αναφερθήκατε προηγουμένως. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προσπαθούμε να αντικατοπτρίσουμε όλες αυτές τις προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, την εκπαίδευση, την βιώσιμη γεωργία, το πόσιμο είδωρ, ε, τις ε, υγειονομικές συνθήκες. Και σίγουρα την φιλετική πολιτική για το φύλλο, ε, που την αναφέρω τελευταία αλλά δεν είναι λιγότερο σημαντική. Έχουμε εργαλεία για να παρακολουθούμε το στοιχείο του φίλου, Προσπαθούμε να είναι όσο δυνατό πιο παρόν στα προγράμματά μας. Γνωρίζετε την προ... τις, πρωτοβουλίες μας, την πρωτοβουλία Spotlight. Πάντως το ζήτημα του φίλου σίγουρα βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας παντού. παρακολουθούμε όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες, για παράδειγμα στο πλαίσιο του Global Aid Fund κλπ. Και προσπαθούμε να εντοπίσουμε οποιασδήποτε καινούριε πρωτοβουλίες εμφανίζονται. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λαμβάνουμε υπόψη αυτές τις προτεραιότητες και οπωσδήποτε για να διατηρήσουμε τα κονδύλια του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Όπως άλλωστε μας επιβάλλεται από τις ε, νομικές μας υποχρεώσεις, ε, από τη νομική βάση επί της εργαζόμαστε. Οπότε συμφωνούμε 100% ε, με την πρόταση που έγινε για αυτό το θέμα. Θέλουμε και εσείς να μας στηρίξετε σε αυτή την προσπάθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα ζητήματα για νούμερα του προπολογισμού του 2019. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε σημαντική αύξηση των πόρων για τη Μέση Ανατολή. 133% αναφέρθηκε πολύ σωστά το ποσοστό αυτό. Αυτό είναι η συνέπεια της απόφασης να χρησιμοποιήσουμε το μη γεωγραφικά προσδιορισμένο απόθεμα. Υπήρχε λοιπόν ένα απόθεμα το οποίο θα μπορούσαμε να το διανύμουμε όπου θέλουμε. Αυτό ήταν επιλογή στην ενδιάμεση ε, αξιολόγηση των προγραμμάτων. Αποφασίσαμε δηλαδή να αυξήσουμε πολύ τις παροχές ε, στην Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα Ιράν, Ιράκ και η Εντό των χωρών τα οποία καλύπτουν, οι οποίες καλύπτονται από το DCI, από το Μηχανισμό Χρηματοδότησης Αναψυχιακής Συνεργασίας, Αυτέ είναι οι χώρε οι οποίε έχουν τι μεγαλύτερε ανάγκε. οι χώρε τη Μέση Ανατολή, η Εμένη, η Ιράν, η Ιράκ. Γι' αυτό το λόγο δώσαμε προτεραιότητα σε αυτέ τι γραμμές του προπολογισμού και σε αυτέ θα χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο τμήμα του Μπορώ να σα δώσω και περισσότερε λεπτομέρειε, περισσότερα στοιχεία αν θέλετε. σχεδόν το σύνολο του αποθέματος το διανέμουμε σε αυτές τις χώρες. Εδώ θα τελειώσω, δεν ξέρω αν ο συνάδελφος από την DG, από τη Γενική Διανύση ΕΚΟ, θέλει να προσθέσει κάτι σε σχέση με τα υπόλοιπα ζητήματα. για το τελευταίο σας σχόλιο για τη Μέση Ανατολή. Εδώ μιλάμε για χρηματοδότηση από το DCI. Πώς θα χρηματοδοτήσουμε δράση στην Ιεμένη με το DCI. Ε, θα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ποσά για αναπτυξιακή βοήθεια πραγματικά. Δεν θα βγούμε εκτός του πεδίου ε, του χρηματοδοτικού οργάνου. να δούμε τις λεπτομέρειες αν θέλετε. Θα σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς θα χρηματοδοτήσουμε με αυτά τα ποσά. Σίγουρα όμως θα εστιάσουμε σε ό,τι είναι δυνατόν να γίνει εντός του πλαισίου του μηχανισμού χρηματοδότησης. Και βέβαια σε σχέση με τους γενικότερους στόχους ανάπτυξης που σχετίζονται με αυτή τη δράση. Δεν πρόκειται να διαφύγουμε από αυτό το πλαίσιο και να χρηματοδοτήσουμε δράσει άλλων οργάνων και μηχανισμών. Λέω στην Ιεμένη δεν μπορούμε να στείλουμε ούτε ε, επίγουσα ανθρωπιστική βοήθεια. Πώ θα χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει. Οι συνάδελφοι θα ζητήσουν λεπτόμερη πληροφόρηση, φαντάζομαι, για το πού ακριβώ θα ε, διανεμηθούν και διατεθούν αυτά τα κονδύλια, τα παραπάνω κονδύλια για τη Μέση Ανατολή, γιατί ε, έχουμε, για παράδειγμα, έλλειψη κονδυλίων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες της Αφρικής. Τέλος πάντων, η Κομισιόν ελπίζω θα μας ε, δώσει λεπτομέρειες, έτσι ώστε τα, μέλη, τα μέλη μας να ενημερωθούν. Γενική Διεύθυνση Ο κύριος Πέρεθ. Ωραία. Ευχαριστώ. Η Γενική θέλει να ευχαριστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την στήριξή του ε, στην επεξεργασία του σχεδίου προπολογισμού 2019. Ε, οι ανάγκε όλο και αυξάνονται, οπότε αυτός ο προπολογισμό αντικατοπτρίζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωση ω σημαντικός δωρητή ανθρωπιστική βοήθεια προσπα... Ε, εξακολουθούν να είμαστε ουδέτεροι, ανθρωπιστές, είναι οι βασικές αρχές, ε, ανεξάρτητοι ε, και αμερόληπτοι. Η... Το σχέδιο προπολισμού 2019 έχει φτάσει στο 1,6 δισεκατομμύριο ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων και 50 εκατομμύριων για να είμαστε έτοιμοι για καταστροφές. Σε ό,τι αφορά τι γεωγραφικές προτεραιότητες, έχουμε Μέση Ανατολή και τις χώρες της γειτονίας συμπεριλαμβανομένης και του, και του, και του Λιβάνου, αυτές που, ε, την Ιεμένη και την Παλαιστίνη. Ε, άλλη γεωγραφική προτεραιότητα η Αφρική, ιδιαίτερα περιοχή του Σαχέλ, ε, το κέρας της Αφρικής και οι μεγάλες λίμνες. Άλλες χώρες και περιφέρειες στις οποίες θα εστιάσουμε είναι το Αφγανιστάν, η Λιβύη και η κρίση Ροχίνγκα. Η εκπαίδευση και η έκταξη καταστάσει είναι ψηλά στην ατζέντα μα. 10% των, του συνολικού προπολογισμού σκοπεύουμε να το διαθέσουμε σε αυτέ. Περιμένουμε ότι θα στείλουμε έτσι ένα ισχυρό μήνυμα στους άλλους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλουμε να είμαστε ηγέτες στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είπατε πως ανέβηκε κατά 10% ε, η χρηματοδότηση για την ε, εκπαίδευση σε εποχές εκτακτής ανάγκης. Έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Τεζουά? Άρνε, ναι. θα θέλατε να προσθέσετε κάτι? Ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι είμαι ε, ευγνώμων για την στήριξη που μου δείχνουν οι συνάδελφοι, ιδιαίτερα εσείς κύριε Ρουμπίκαλα, καλά και ε, χαίρομαι επίσης που η κυρία Χάουταλα τόνισε το θέμα της ε, διατύπωσης, ε, των ελλείψεων που υπάρχουν λίγο στη διατύπωση. Νομίζω πως πρέπει να γίνει λόγος για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και χαίρομαι πολύ που δεν είμαι μόνος σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να ε, συντονίσουν τις θέσεις τους. Όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, η συζήτηση θα γίνει αύριο. Όμως ε, θα θέλα να πω ότι θα θέλαμε να τονίσουμε τις πτυχές της εκπαίδευσης, της ε, εκπαίδευσης ιδιαίτερα σε, εποχές, σε περίοδους κρίσης και στην διάσταση του φίλου, στις γυναίκες. Πρέπει να καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες για ενίσχυση της θέσης των γυναικών. αλλά και στο σημείο 3α πρέπει να δοθεί βάση για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να επανέλθω τώρα στο ότι φυσικά και η ανθρωπιστική βοήθεια ε, δεν είναι αναπτυξιακή βοήθεια, δεν είναι το ίδιο πράγμα, πρέπει να υπάρξει ένας αφής διαχωρισμός. Και επίσης θα χρειαστεί να κοιτάξουμε τις λεπτομέρειες ε, των γειτονικών χωρών έτσι ώστε να μην ε, αφήσουμε κανέναν πίσω. Αλλά να εξετάσουμε και με προσοχή τις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού, να δούμε πού διοχετεύονται κονδύλια και ε, για να διευκρινίσω κάτι Ε, να ευχαριστήσω καταρχά ε, τον Έσαλ και την αναφορά του στο Brexit. Να πω εδώ ότι, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια χώρα η οποία έχει δεσμευτεί για το 0,7%. Μας είπατε και πως ε, πρέπει να συμπεριληφθεί και το κόστος των ε, προσφύγων ε, στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Η Γερμανία το έχει τονίσει, όμως εγώ θεωρώ πως αυτό πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και πως είναι εθνικό θέμα. Όμως άμα δεν ε, ξεκινήσει μια συζήτηση για το τι μπορούμε να δεχτούμε και τι όχι, τι είναι αποδεκτό γενικά και τι όχι, τότε νομίζω πως θα κρυβόμαστε πίσω από αυτή τη γραμμή του προπολογισμού και θα το χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για διάφορες ε, στάσεις. Μα αναφέρθηκε επίσης και το καταπίστευμα για την Αφρική, το ποσοστό αυτού. Ας είμαστε λοιπόν σαφείς και συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Ας δούμε μία-μία την κάθε γραμμή του προϋπολογισμού και ας δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη ξεχωριστά για την αναπτυξιακή βοήθεια. Και ο Σάιλ στο τελευταίο ψήφισμα μας ε, τονίζει ότι το 0,7% είναι ένα νούμερο που πρέπει να ε, μην ξεχνάμε, να το επαναλαμβάνουμε διαρκώς. Αυτά από μένα προς το παρόν. Αυτές είναι οι σκέψεις μου μέχρι στιγμής. Ελπίζω να συνεργαστούμε καλά και να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα για τη θέση μας και να αποτελέσει αυτό αφετηρία περαιτέρω συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κρατημέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σαρλ και Χέντι, θέλετε να προσθέσετε κάτι. ξέχασα κάτι. Στο πλαίσιο του διαρθωμένου διαλόγου είχαμε αναφέρει στο πλαίσιο της, των ενδιάμεσων εκθέσεων. Ε, είχα ρωτήσει την Κομισιόν, τους εκπροσώπους εξωτερικής δράσης, τι γίνεται με την εφαρμογή της αρχής της διάκρισης. Η απάντηση ήταν ε, αόριστη. Αλλά όταν έγινε στο Στρασβούργο η συζήτηση με την κυρία Μογκερίνη και τον Επίτροπο Μιμίτσα, είναι, έγινε σαφές ότι αυτή η αρχή πλέον δεν εφαρμόζεται. Α το πούμε ξεκάθαρα. Γιατί σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, θα πρέπει να ξέρουμε ποιε είναι οι αρχέ που τον διέπουν, που διέπουν τη δημοσιονομική μα πολιτική. Τότε είχαμε δώσει ένα αγώνα. Αν τώρα αυτή η αρχή δεν ισχύει πλέον, α το πούμε. Υπάρχουν πλέον επιχειρήματα λοιπόν για να μην εφαρμόζεται αυτή η αρχή. Αν θέλουμε να έχουμε στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τους φτωχούς των λιγότερων επιτυγμένων χωρών και αν η αρχή της ε, διάκρισης, της διαφοροποίησης δεν λειτουργεί πια θα πρέπει να το πούμε. Το βλέπουμε βέβαια στα νούμερα, αλλά θα ήθελα να μας εξηγηθεί κιόλας. Γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια η, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης αφενός και το κοινοβούλιο αφετέρου είχαν ξεκινήσει διαφορετικά. Ε, ε, χώρες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα ε, έχουν πολλές φορές καταστραφεί από τις σειράξεις και τώρα προσπαθούμε να τις οικοδομήσουμε πράγματι. Ε, κυρία Χάουταλα, ε, η ασφάλεια και μετανάστευση είναι δύο πτυχές στις οποίες θα πρέπει να τις προσέχουμε πάρα πολύ να μην ξεκινήσουμε ε, και διαχέουμε την αναπτυξιακή βοήθεια σε άλλους στόχους που δεν έχουν σχέση ή και έρχονται σε αντίθεση με την ανάπτυξη. Η Κομισιόν ανέφερε την πρωτοβουλία Spotlight. Τη στηρίζουμε προφανώς. Ενώ για την ανθρωπιστική βοήθεια μας είπε η Κομισιόν ότι ένας από τους στόχους τώρα είναι να στηρίξουμε μια λύση για την κρίση των Ροχίνγκα Εκεί έχουμε βιασμένε γυναίκες, τεράστια ανθρωπιστική κρίση. 65.000 γυναίκες έχουν ήδη γεννήσει ή θα γεννήσουν ένα παιδί που είναι αποτέλεσμα των μαζικών ομαδικών ε, βιασμών στην ε, Μιανμάρ. Παρακολουθεί η Κομισιόν αυτό το θέμα. Είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο σεξουαλικής ε, βίας στα χρονικά. Και η Αυστριακή Υπουργός θα έρθει να μα ενημερώσει, οπότε μπορούμε να τη ρωτήσουμε. Τώρα δεν ξέρω αν η Κομισιόν, η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ μπορεί να μα πει ότι αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ειδικά για αυτέ τι γυναίκε που είναι θύματα εξουσιαλική βίας. Δεν γνωρίζω, θα σα απαντήσω κάποια άλλη στιγμή. Ωραία, θα ρωτήσουμε το Συμβούλιο. στι 11 θα είναι εδώ ο υπουργό. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Θα πρέπει να ελέγξουμε πού πηγαίνουν τα χρήματα, θα ενημερώσουμε τα καινούργια χρηματοδοτικά όργανα τροπολογίες μέχρι τις 18 Ιουλίου το μεσημέρι, την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Okay, thank you. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 8 τώρα. Η νέα συμμαχία για την επισητιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Μετά από την έκθεση, δηλαδή συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Μαρία Χόιμποκ πριν από δύο χρόνια έχει περάσει, έχουν περάσει ήδη δύο χρόνια. Τρέχει ο χρόνος. Θα μας ενημερώσει λοιπόν για το USG 8 και θα μας πει για την πρωτοβουλία που ξεκίνησε όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις στον αγροτροφικό κλάδο. Το θέμα είναι τι έγινε αυτά τα δύο χρόνια. Θα ακούσουμε κάποιους εμπειρογνώμονες λίγο από την Αφρικανική Ένωση. Έχουμε εδώ τους προσκεκλημένους μας και από την δράση κατά της πείνας. Μαρία, θέλεις να κάνεις μια εισαγωγή γιατί κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα και τι διακυδεύεται ακριβώς που πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Λίγα λεπτά για εξήγησέ μας. Σας ευχαριστώ πολύ Λίντα. Ναι, λοιπόν, γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί καταρχάς το θέμα αυτό με απασχολεί πάρα πολύ. Το θέμα της γεωργίας στην Αφρική και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες είναι κάτι που πρέπει να προβληθεί. Χρειάζεται ε, βοήθεια διότι η στάση απέναντι στην καινοτομία είναι εχθρική μάλλον θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν είναι επίγουσα ανάγκη να αλλάξει κάτι και για μένα αυτό αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε ε, την πείνα πρέπει να αρχίσουμε από τη γεωργία, από τους αγρότες. Και αφετηρία και αρχή των επενδύσεων ε, είναι όχι να δίνουμε τα λεφτά στο χέρι, αλλά να χρηματοδοτούμε στοχευμένα σε συγκεκριμένα επιλεγμένα καλά έργα τα οποία θα στηρίζουν τους ε, μικρούς αγρότες, ε, γιατί αυτοί οι αγρότες ε, είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας. Στην υποσαχάρη Αφρική το 60% των κατοίκων ζει, στις, ζει στην Ήπεθρο, σε αγροτικές περιοχές. Το New Alliance είναι και ο λόγος για τον οποίο ασχολούμαι με την έκθεση αυτή. Δεν είναι business as usual, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ε, χρησιμοποιεί επιχειρηματικά μοντέλα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ε, συνα άδει με τους στόχους ε, του 2030 και ε, προσπαθεί να ενημερώσει και να συλλέξει ταυτόχρονα πληροφορίες για την κατάσταση της γεωργίας εκεί. Με, έχουμε συνεργαστεί με τον Παγκόσμιο Επιστημικό ε, Οργανισμό με εκπροσώπους από όλον τον κόσμο σε συνέδρια έτσι ώστε να συζητηθούν αυτά τα θέματα. Και το περασμένο Σαββατοκύριακο ήμουν στην Κρήτη όπου συναντήθηκαν επιστήμονες από όλο τον ε, κόσμο για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψει σχετικά με τις διάφορες ε, νέες ε, τεχνολογίες και μεθόδους γεωργίας. Η New Alliance λοιπόν ε, συμμετέχει ενεργά σε όλες αυτές τις προσπάθειες. Προσπαθούμε να αντλήσουμε διδάγματα, να βγάλουμε, να συλλέξουμε τις βέλτιστες πρακτικές έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσουμε για το σκοπό της ε, στοχευμένης πλέον στο μέλλον χρηματοδότησης και της στήριξης των μικρών αγροτών. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τους πόρους μας. Αυτά λοιπόν από μένα προς το παρόν και χαίρομαι πολύ για την ε, ερχόμενη απόψεων. Σας ευχαριστώ. Η πρώτη παρέμβαση που θα έχουμε θα είναι μέσω Skype. Δεν θα υπάρξει όμως ε, διερμηνία, θα είναι στα αγγλικά, επειδή η ποιότητα μπορεί να είναι προβληματική. Μαζί μας λοιπόν θα έχουμε, και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, τον κύριο Ουσμάν Μπαντιάνα από το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για τις Επισητιστικές Πολιτικές. Έχει εκπονήσει μια αξιολόγηση ποιότητα εκ μέρου τη Αφρικανική Ένωσης. Είσαστε εδώ, κύριε Μπαντιάν. Καλώς ήρθατε μέσω Skype στην Επιτροπή μας. Δεν ξέρω πού βρισκόσαστε όμως. Μπορείτε και να μας πείτε από πού είσαστε. Thank you very much. I give you the floor. Okay, thank you, ma'am. I am actually calling in today from Lilongwe in Malawi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 Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν για την ε, παρουσίασή σας. Βλέπω πως έχετε πολλές ε, εκδηλώσεις προγραμματίζετε με συμμετοχή των δωρητών, οπότε αυτά όλα είναι πολύ θετικά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Βαλαντάν Ροσάρ από την Action Against Hunger και θα μας ε, μιλήσει στη γλώσσα του. Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Είμαι υπεύθυνο για την επισητιστική βοήθεια και για την καταπολέμηση της ε, φτώχειας. Εγώ θα υπογραμμίσω την άποψη της κοινωνίας των πολιτών και των ε, παραγωγών τροφίμων σε σχέση με αυτή τη νέα συμμαχία για την επισητιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπενθυμίσω ότι ξεκινήσαμε το 2012. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία βέβαια έγινε ευπρόσδεκτη γιατί κατέληξε μετά από 30 χρόνια που δεν δίναμε προτεραιότητα στην αγροτική ανάπτυξη και τον επισητιστικό κλάδο, επιτέλους έγινε. Οπότε ξαναβάλαμε τα θέματα που είχαν να κάνουν με την διατροφή, κάτι που περιμέναμε πολλά χρόνια. Όμως τόσο όσον αφορά τη μορφή, όσον αφορά και την ουσία και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η πρωτοβουλία αυτή, πέρασε από πολλές επικρίσεις και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές αδυναμίες οι οποίες επηρέασαν τον αντίκτυπό της. Και εδώ θα αναφερθώ στις κύριες τρεις αδυναμίες που, με τις οποίες συμφωνούν οι περισσότερες οργανώσεις παραγωγών της υποσαχάριας Αφρικής αλλά και πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Από την αρχή, από το 2012, είπαμε ότι δεν βοηθάει τη συμμετοχή όλων. Ήταν μια πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της, ε, του λοιμού, της κακής διατροφής κτλ. Αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες οργανώσεις που ασχολούνται με αυτό το θέμα, ούτε όταν δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία αυτή, ούτε και στην υλοποίησή της. Για παράδειγμα, στάλει ανοιχτή επιστολή από μια οργάνωση στην οποία συμμετέχουν ε, όλες οι οργανώσεις παραγωγών τη Δυτικής Αφρικής. Το 2012 έγινε αυτό, πήγε στην Αφρικανική Ένωση. Ήταν ανοιχτή επιστολή, άρα μπορεί κανείς ε, να τη δει. Και λέει ότι ο περισσότερος πληθυσμός ε, ασχολείται με την γεωργία, αλλά το 80% της παραγωγής δεν φτάνει στον προορισμό της. Οπότε τελικά ήταν περίεργο πως μια πρωτοβουλία η οποία είχε σαν στόχο να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις για να καταπολεμηθεί η έλλειψη διατροφής δεν ελήφθη υπόψη. Μια άλλη κριτική που έχουμε να κάνουμε αφορά περισσότερο την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Αν δούμε τι έγινε στην Ποσαχάρια Αφρική με την πρωτοβουλία αυτή, διαρθρώνεται γύρω από ανάγκες, που όμως δεν είναι οι ανάγκες των μικρών ε, αγροτών ε, ή των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Οι περισσότερες επικρίσεις που έγιναν από διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις παραγωγών έχουν να κάνουν με το στρατηγικό πλαίσιο επειδή διαρθρώνονται γύρω από τις ανάγκες των πιο μεγάλων επιχειρήσεων και των διεθνών ομίλων αγροτροφικού τομέα. Και λένε ότι σε πολλές περιπτώσεις το πλαίσιο στρατηγικής το οποίο κατεύθυνε και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας δεν έβαλε, έλαβε υπόψη τις ε, ανάγκες των πιο μικρών. Κατά τη γνώμη μου, το ότι δεν ε, λήφθησαν υπόψη οι μικρή παραγωγοί οφείλεται στο ότι δεν συμμετείχαν από την αρχή. Δεν ήταν παρόντες στη συζήτηση, δεν ήταν παρόντες στην Επιτροπή Κατευθυντήριων Γραμμών, οπότε δεν μπόρεσαν να εκφράσουν την άποψή τους και να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Όμως για μένα τίθεται το ζήτημα αυτή η νέα συμμαχία για την επισητιστική ασφάλεια και τη διατροφή, πού προορίζεται, για ποιον έχει φτιαχτεί, τα άτομα αυτά λοιπόν που αποτελούν το 80% της κοινωνίας στην Αφρική δεν ε, μπόρεσαν να πούν τη γνώμη τους. Ποιοι λοιπόν επωφελούνται κύριοι από τη Νέα Συμμαχία. Αυτό είναι ένα ερώτημα που θέτουν πολλοί και στην οργάνωση των Αφρικανών παραγωγών αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς. Η τρίτη αδυναμία, η τρίτη κριτική που έχουμε να εκφράσουμε είναι οι πραγματικές επιπτώσεις της νέας αυτής συμμαχίας για την επισητιστική ασφάλεια και την διατροφή. Είναι δύσκολο να μετρηθεί βέβαια και δεν μετριέται. Υπάρχει πρόβλημα δικτών. Οι δίκτες είναι πάρα πολύ γενικοί. Είναι δίκτες που δεν είναι συγκεκριμένοι, δεν είναι δείκτες επιπτώσεων και αυτό για πολλούς λόγους. Σε μερικές περιπτώσεις Τότε βέβαια δεν συμμετείχα εγώ στις συζητήσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει υποθεί ότι οι δείκτες αυτοί επιπτώσεων για τις επενδύσεις τέθηκαν στο τραπέζι, αλλά θεωρήθηκαν πάρα πολύ αυστηροί, τρόμαξαν ουσιαστικά τις ιδιωτικές επενδύσεις. Οπότε τίθεται το ζήτημα αυτό των δικτών, αλλά τίθεται και το θέμα και των Ε, βασικών ε, στοιχείων της πρωτοβουλίας. Ότι δηλαδή αυξάνοντας τις επενδύσεις αυτόματα θα έχουμε περισσότερη επιστηστική ασφάλεια. Όμως αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλοϊκό, αυτή η σύνδεση που γίνεται. Γιατί η επιστηστική ανασφάλεια και η κακή διατροφή έχουν ε, βαθιές αιτίε που είναι διαρθρωτικές, που έχουν να κάνουν με θέματα ισότητας, με θέματα πρόσβασης, με την φτώχεια και δεν αντιμετωπίστηκαν από τις χώρες που συμμετέχουν στην εκπόνηση του στρατηγικού πλαισίου. Όμως είναι και θέμα κατανόησης της πραγματικότητας όσον αφορά την επιστημιστική ανασφάλεια στην υποσαχαρή Αφρική. Αν περιοριστεί η παραγωγή. Ξεχνάμε πάντα το θέμα της πρόσβασης. Είτε της ε, πρόσβασης ε, της φυσικής, πώς να φτάσει κανείς στα τρόφιμα, ή και το θέμα των πόρων. Όλοι λένε ότι πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή τροφίμων. Το θέμα είναι όμως πώς και ποιος θα υποφεληθεί από αυτήν. Και ένας, ε, μια από τις ε, αιτίες που αναφέρει η κοινωνία των ε, πολιτών όσον αφορά τις λίγες συνέπειες που τελικά έχει νέα συμμαχία στην καταπολέμηση της επιστημικής ανασφάλειας είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε ένα αγροτικό μοντέλο το οποίο δεν είναι βιώσιμο, δεν θεωρούμε βιώσιμο είναι ένα μοντέλο που δεν λαμβάνει υπόψη επαρκώς το τι θέλει και τι ζητά ο κόσμος, ποιες είναι οι ανάγκες του, ούτε λαμβάνει υπόψη επαρκώς την κλιματική αλλαγή που διπλασιάζει τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή στην Αφρική από ό,τι στην Ευρώπη. Συνεπώς έχουμε μια νέα συμμαχία που μετά το 2012 που ξεκίνησε δεν έχει τις επιπτώσεις που να μπορούμε να μετρήσουμε όσον αφορά την επισητιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Υπάρχουν βέβαια κάποια προγράμματα που μπορούν να προωθηθούν, που όντως στόχευσαν τους μικρούς παραγωγούς και την πρόσβαση στην αγορά, πράγματι. Αλλά αυτά είναι λίγα και δεν φτάνουν. Θα πρέπει να υπάρχουν άλλα προγράμματα, πιο μεγάλα. Στην ε, Νιγηρία, στη Μπουρκίνα Φάσο είχαν αρνητικές συνέπειες και οδήγησαν σε κάποια μοντέλα ανάπτυξης που τελικά μείωσαν τα έσοδα των αγροτών από τις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις. Αυτές είναι οι τρεις κύριες ανησυχίες. Η κριτική δηλαδή που επιφέρουν η παραγωγή και η κοινωνία των πολιτών κάπου 100 μη κυβερνητικέ οργανώσεις και παραγωγή κατέληξαν σε αυτές τις αδυναμίες και κάναμε και μελέτες σε 6-7 χώρες, η Κένια, Μαλαουή, Μπουργίνα Φάσο, ε, Σενεγάλη, Ακτή Λεφαντοστού, που συμμετέχουν στη Νέα Συμμαχία. Και όλες αυτές οι επικρίσεις υπάρχουν ε, και στις συστάσεις και στα αποτελέσματα των τεσσάρων μελετών που αναφέρθηκαν ε, πριν στην παρουσίαση που ακούσαμε. Θα αναφερθώ σε δύο τώρα συγκεκριμένε περιπτώσει από μελέτες που έκανε στην Υπουργένα Φάσο η Γαλλία και που περιλαμβάνουν τα τρία σημεία, τι τρεις ανησυχίε που σας ανέφερα και εγώ για το ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, τι επιπτώσεις έχει και ποιος επωφελείται και εξού και η Γαλλία εγκατέλειψε τη Νέα Συμμαχία Κάπως ε, μονόπλευρα μεν το αποφάσισε, αλλά το αποφάσισε ακριβώς γιατί το μοντέλο χρηματοδότησης και ανάπτυξης που προτείνει δεν αντιστοιχεί στην αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης της επισητιστικής ανασφάλειας και της κακής διατροφής. Οπότε κάνω έκκληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αυτή συμμαχία ήταν συντονιστής στην ακτή Ελεφαντοστού. Και όταν μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφυγε από τη Νέα Συμμαχία και τρεις χώρες έκαναν μελέτες επιπτώσεων που δείχνουν ότι οι επιπτώσεις δεν είναι τόσο θετικές, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της να προβεί σε μία μελέτη αντικτύπου για τις συνέπειες και τις επιπτώσεις του μοντέλου της νέας συμμαχίας στην επιστηστική ασφάλεια και τη διατροφή στην ακτή ελεφαντοστού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Έχουμε καθυστερήσει λίγο. Ε, η υπουργό θα έρθει πολύ σύντομα. Η συζήτηση για τον προπολογισμό μας πήρε πιο πολύ χρόνο από ό,τι θέλαμε. Οι Γάλλοι από την άλλη μεριά μας λέγατε, μας είπατε, «εγκατέλψαν τη συμμαχία. Ε, παρόλο που ε, έχουμε νέα και για κάποιες επιτυχίες της συμμαχίας. Μαρία, θες να πεις δύο λόγια και μετά θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ναι, πολλές ερωτήσεις έχω βασικά. Όμως ε, πρέπει να περιοριστώ, διότι δεν έχουμε και χρόνο. με ενδιαφέρει για αυτούς που θα κάνουν τις αξιολογήσεις πώς ε, αυτό συνδέεται με το θεματολόγιο του 2020. Θα υπάρχει αξιολόγηση και αυτού. Μετά, οι ίδιοι οι αγρότες έχουν συμμετάσχει στην ε, διαδικασία. Ε, το λέω αυτό πάνω σε αυτό που είπατε εσείς για, την, για το ποσοστό συμμετοχής, ότι δεν χρησιμοποίησαμε τη γνώση τους κτλ. Μια λοιπόν που αναφέρεστε σε αυτήν την αξιολόγηση, τι γίνεται με θέματα όπως η βιοπικιλότητα, η πρόσβαση στη γη για τους αγρότες, για τους πολίτες εκεί που ζουν εκεί. Και ε, μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι συμπεράσματα εξάγεται από αυτήν την αξιολόγηση Ακριβώς διότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα επενδύσεων ε, γεωργικών, το EIP. Τι μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε και πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτόν τον τομεακό διάλογο με τις χώρες εταίρους να προσφέρει νέες ε, μεθόδους ε, καλλιέργειας, γεωργίας για την ε, βελτίωση της κατάστασης εκεί, αν υπάρχουν κάποιες προτάσεις για βιολογική γεωργία, τι μπορείτε να μας πείτε. και επίσης ε, πώς είναι η συνεργασία σας ε, με τους διάφορους άλλους οργανισμούς έτσι ώστε να ανταλλάξετε τις πρακτικές. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε δίκιο. Το Ταμείο βιώσιμη ανάπτυξη. θα δώσει, ε, στη συζήτηση μάλλον για το Ταμείο βιώσιμη Ανάπτυξης θα δοθεί έμφαση σε αυτά που αναφέρατε. Είναι λοιπόν μια προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν, ποιες είναι οι δικέ σας εκτιμήσεις για αυτές τις νέες ε, γραμμές του προπολογισμού, τις επενδύσεις. Γιατί δυσαρεστήθηκε η Γαλλία, τι συνέβη. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των ιδιωτικών επενδύσεων στη Γεωργία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Νέα Συμμαχία, ήταν μια δικασία που είχε ξεκινήσει, ξεκινήσει από το G8 πριν από 6 χρόνια. Ε, ξεκίνησε στη Λαλάκυλα της Ιταλίας ε, και η διαπίστωση ήταν ότι γινόντουσαν πολύ χαμηλές ε, το οποίο των επενδύσεων ήταν πολύ χαμηλό Επίσης έχουμε την, το GAPS, το παγκόσμιο πρόγραμμα για την ασφάλεια των τροφίμων. Από εκεί ξεκίνησε λοιπόν. η Γάλλη αποσύρθηκαν μονομερός. Γνωρίζουμε ότι αν κανείς δει το site της ε, Νέας Συμμαχίας θα διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση. Δεν δείχνει εδώ και τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια να έχει κάποια δραστηριότητα. Ε, το γνωρίζουμε αυτό. Μπορούμε να κάνουμε αξιολογήσεις, το είδαμε, ας πούμε, ακούσαμε την, την, ε, το IFPRI, την ε, ε, παρουσίαση του ΙΦΠΡΙ. Γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά τα σχόλια, αυτές τις κριτικές. θέλουμε να εξασφαλίσουμε βιοπικιλότητα, καλή διατροφή, διαφάνεια στις τιμές λοιπά Και χρειάζεται να εντείνουμε την εστίασή μας στην, ε, στο θέμα των τροφίμων. Το δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε προβλέψει μέχρι το 2020 στο, για, το, για το θέμα αυτό. Ε, ξετάζουμε όμως ε, με καινούριο τρόπο το ιδιωτικό τομέα χωρίς να τον περιορίζουμε σε μια διαδικασία G8 ή νέα συμμαχία. Παρόλο ότι η διαδικασία του G8 ε, παρακολουθείται ακόμα από πλευρά λογοδοσία. Τώρα, για τα εναλλακτικά συστήματα και το EIP, ε, που γίναν δύο ερωτήσει. Υπάρχει ακόμα πολλή αντίδραση, έλλειψη ενθουσιασμού, να το πω έτσι, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να επενδύσουν σε τρόφιμα και γεωργία. Γίνονται πολλές επενδύσεις στις πόλεις, στις αστικές περιοχές, στη ψηφιοποίηση και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, λιγότερο στις ε, αγροτικές εκμετάλλευσει και τη γεωργία. Είναι πιο υψηλός ο κίνδυνος, ε, γι' αυτό το λόγο το αποφεύγουν. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και να δούμε και τα αίτια βέβαια. Τους τελευταίους μήνες εξετάσαμε διάφορες πρωτοβουλίες μέσω των οποίων θα μπορούσαμε να δώσουμε απάντηση στα όσα έχουμε ήδη συζητήσει. Με το, ε, έχουμε 20 εκατομμύρια ήδη επενδύσεις σε μικροδάνεια. Αποκινούμε τον ΦΑΟ επίσης σε χαμηλό επίπεδο χρηματοδοτούμε ε, με ποσά 20.000 μέχρι 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ε, τα πιο χαμηλά από ό,τι συνήθως που ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο. ...39 εκατομμύρια με τον FMO και 30 εκατομμύρια με την KFW. Έχουμε ένα συνολικό ε, ποσό ε, χαρτοφυλάκιο 134 εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να παρακολουθούμε όλα αυτά βέβαια τα οποία τρέχουν μέσα με αυτό το ποσό και να τα αξιολογούμε. Είναι σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις επιτόπου. Τι μοντέλα χρησιμοποιούμε. Ε, ε τα είπαμε στη Ρώμη πριν από μερικούς μήνες αυτά. Σύμφωνα με τι εμπειρίε μα έχουμε καταλήξει τα εξή συμπέρασματα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να συνεργαστούμε με τον ιδιωτικό τομέα σε ό,τι αφορά τι διαδικασίες μεταρρύθμισης του τομέα των τροφίμων. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνική συνδρομή και το ε, ρυθμιστικό περιβάλλον και το EIP. E ε, πρέπει να βρούμε το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο για να βοηθήσουμε τις επενδύσεις. Και δεν μιλώ μόνο για ευρωπαϊκές επενδύσεις γιατί έχουμε τη διαδικασία της, ε, των βιώσιμων ε, επιχειρήσεων στην Αφρική. Ε, με τη Γενική Διεύθυνση Άγκρη προσπαθούμε να εντοπίσουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να εμπλέξουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη και το κλιματολογικό και το κοινωνικό ε, ένα μοντέλο δηλαδή που θα συνδυάζει την οικονομία με, την, ε, με τις κοινωνικές και επιβαλλοντικές πτυχές και ιδιωτικές επενδύσεις ε, στην, ανάπτυξη, στην έρευνα και την ανάπτυξη. Χρειάζεται περισσότερε, χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα. Βιοποικιλότητα, αγροδασοκομεία, ε, διαφοροποίηση στα τρόφιμα τα οποία χρησιμοποιούνται για την ανθρώπινη κατανάλωση κλπ. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μία προσέγγιση της ε, βιομηχανίας τροφίμων ε, την οποία προσέγγιση όμως θα υιοθετήσουν οι χώρες της Αφρικής και που θα βάζει ψηλά στην ατζέντα την επενδύσει στα τρόφιμα, το μέτρο τροφίμων και σε επιχειρήσεις σχετικές. Χρειαζόμαστε όμως και μια καινούργια διακυβέρνηση. Η Επιτροπή για την ε, Τροφιμική Ασφάλεια, για παράδειγμα, θα πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή αυτής της διακυβέρνησης. Το, ο τύπος των συστημάτων τροφίμων τι επόμενε δεκαετίες θα είναι πολύ διαφορετικός, ιδιαίτερα με την Ατζέντα 2030. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει και στο Συμβούλιο Στρατηγικής, έτσι. Δεν συζητήσαμε πώς ακριβώς θα μπορούν οι επενδύσεις στρατηγικά μιλώντας να βοηθήσουν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 ξέρω την ε, περίπτωση της Βουρκίνα Φάσο μόνο, οπότε η... υπήρξε διαβούλευση για τις επιπτώσεις της νέας συμμαχίας ε, στις ζωές τους. Το ΣΥΡΑΤ που είναι ένα ερευνητικό κέντρο έκανε μια μελέτη με αυστηρή μεθοδολογία και προσπάθησε όντως να έχει σε επαφέ με όλους τους ενδιαφερόμενους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Πρέπει να κλείσουμε εδώ αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε από τόσο μακριά για να είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπροσά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα παρακολουθούμε αυτή την υπόθεση και θα φροντίσουμε όταν επενδύουμε σε νέους μηχανισμούς να σκεφτόμαστε καλύτερα πριν. Ωραία, κλείνει αυτό το θέμα. Και τώρα, περιμένουμε την Προεδρία, την Αυστριακή Προεδρία. Okay, colleagues. We, if everyone could... Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ να καθίσετε, διότι έρχεται ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της συνεδρίασής μας. Βρίσκεται εδώ η υπουργό εκ μέρους της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου. Έχουμε λοιπόν την τιμή να υποδεχτούμε την κυρία Καρίν Κνάισελ, Α, μάλιστα βλέπω Κνάισελ, σας λένε εγώ το πρόφερα λάθος. Ε, Υπουργό για Ευρωπαϊκά Ζητήματα, Ενσωμάτωση και Εσωτερικές Υποθέσεις. Με μεγάλη μας χαρά λοιπόν σας υποδεχόμαστε σήμερα κύριε Υπουργέ. Οι επόμενοι έξι μήνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί όπως γνωρίζετε κι εσείς. Περνάμε στο τελικό στάδιο της θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στους τελευταίους 9 ή 10 μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Γνωρίζετε επίσης ότι αυτή τη στιγμή διανύουμε έναν αριθμό μεγάλων και σοβαρών ανθρωπιστικών κρίσεων και αυτή η κατάσταση είναι χωρίς προηγούμενο. Οι κρίσεις έχουν ενταθεί, έχουν διευρυνθεί, έχουν μεγαλώσει σε διάρκεια. Υπάρχουν εκτοπισμένοι άνθρωποι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προσπαθούμε να επικεντρωθούμε στην ανθρωπιστική βοήθεια, ιδιαίτερα ε, στα παιδιά. Βλέπω στο βιογραφικό σας ότι έχετε δραστηριοποιηθεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και σας έχει απασχολήσει το θέμα των ε, ανήλικων προσφύγων και στην Τουρκία και στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε για τον ε, προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση στον προϋπολογισμό για ανθρωπιστική βοήθεια. για την ανοικοδόμηση, για την αντιμετώπιση κρίσεων ε, σε χώρους που διανύουν κρίση και την ανοικοδόμηση χωρών που πέρασαν από κρίση. Σας δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί διερμηνείς. Είχα χθε τη χαρά να συνομιλήσω με βουλευτές της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και το λέω και το εννοώ. Η συνεργασία και η συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συγχωρείτε, είστε Μπορείτε να είστε λίγο πιο ησυχοί. Ναι, αν θέλετε να μιλήσετε, όπως το είπα, μπορείτε να το κάνετε εκτός της αίθουσας. Εδώ συνεδριάζουμε. Με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Το θεωρώ λοιπόν τιμή μου που βρίσκομαι εδώ για να ανταλλάξω απόψεις ουσιαστικά μαζί σας με τους ευρωβουλευτές, διότι εσείς βρίσκεστε εδώ για να ελέγχετε εμάς τους εκπροσώπους της ε, Προεδρίας, σε ένα βαθμό εκπροσώπους της εκτελεστικής εξουσίας δηλαδή, και προσβλέπω στην ε, συνεργασία μας, όπως έκανα και το τελευταίο εξάμηνο, επτάμηνο, προετοιμαζόμενοι για την Προεδρία. Ελπίζω λοιπόν να είναι η αφετηρία η σημερινή ανταλλαγή απόψεων για μια πολύ επικοδομητική συνεργασία στο επόμενο εξάμεινο. Θα μιλήσω αγγλικά και γαλλικά και θα αρχίσω λοιπόν από τη γαλλική γλώσσα παραθέτοντας τον Μοντεσκέ ο οποίος αναφέρεται συγκεκριμένα στην ε, ισορροπία δυνάμεων. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, είναι τιμή μου και χαρά μου να σας απευθυνθώ σήμερα ως Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας και προφανώς ως Προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου καταρχήν να σας βεβαιώσω ότι αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ε, είναι μια κοινοβουλευτική συνέλευση όπως άλλων οργαν, οργαν, διεθνών οργανισμών, αλλά είναι η μόνη η οποία ε, εκλέγεται απευθείας από τους ευρωπαϊκούς λαούς. Μία από τις βασικές αρχές της ε, δημοκρατίας στην Ευρώπη είναι η αρχή του διαχωρισμού των εξουσιών, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική. Και χρησιμοποιώντας αυτή την όμορφη γλώσσα του Μολιέρου, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω αυτό που είχε πει ο Μοντεσκιό. Το 1748 έγραφε στο έργο του ο νόμος, το, το, το πνεύμα των νόμων ότι δεν υπάρχει ελευθερία αν η δικαστική εξουσία δεν διαχωρίζεται από την νομοθετική και την εκτελεστική. Και ακόμα πιο κάτω λέει δεν θα είχαμε τίποτε, τίποτα αν ο ίδιος ασκούσε και τις τρεις εξουσίες. Δηλαδή ο ίδιος έκανε τον νόμο, τον εκτελούσε και δίκαζε τα αδικήματα με βάση αυτό τον νόμο. Οπότε θα συνεχίσω στα αγγλικά. Η ουσία λοιπόν της ε, ομιλίας μου είναι πως ε, βρίσκομαι εδώ ενώπιον της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης και εκτιμώ πολύ την ευκαιρία που μου δίνεται να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως σας είπα, έχω αρκετό χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις, διότι εσείς είστε εδώ για να ελέγχετε εμάς. Η Αυστρία λοιπόν Μόλις ανέλαβε την Προεδρία πριν από λίγες μέρες, βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της αναπτυξιακής συνεργασίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία επαναπροσδιορισμού ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας για τα επόμενα ε, χρόνια. Αυτό ως ε, μέρος του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου. Θα μπω όμως στο τέλος της παρουσίασής μου σε αυτό. Επίσης επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση μας με τις χώρες ΑΚΕ στα πλαίσια της ε, αντίστοιχη συμφωνίας. Της συμφωνία δηλαδή του Κοτονού. Και όλα αυτά γίνονται ε, στο πλαίσιο αυξανόμενων συγκρούσεων με ε, αυξανόμενο αντίστοιχα αριθμό προσφύγων. 65 εκατομμύρια πρόσφυγες εκτιμώνται πως υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πλανήτη μας. Ε, γνωρίζετε κι εσείς ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή και οι εσωτερικά εκτοπισμένοι άνθρωποι. Αυτό λοιπόν ε, που αντιμετωπίζουμε ξεπερνά τα όρια της ε, διεθνούς συνεργασία και της ανθρωπιστικής βοήθειας όπως την ξέρουμε τα τελευταία 30 χρόνια. Ωστόσο πρέπει και εμείς και μπορούμε να συνεισφέρουμε με επικοδομητικό τρόπο θα, ακούσω, θα ακούσετε από, μένα την ε, ε, φράση «συνοχή πολιτικής». Είναι κάτι πολυδιάστατο και πρέπει να ε, είναι χαρακτηριστικό της ευρωπαϊκής πολιτικής, ιδιαίτερα ε, με τις σχέσεις της προς Ανατολή και Δύση. Θα σταθώ όμως στην κυριότερη προτεραιότητα η οποία μας ε, απασχολεί από την εποχή των στόχων του Μοντερέι. Είναι δηλαδή η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας και η εξάλληψη αυτής. Στην προηγούμενη μου σταδιοδρομία ως ε, αναλύτρια εξωτερικών σχέσεων έχω γράψει πολλές φορές για το θέμα αυτό και έχω αναφερθεί πολλές φορές στην προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ότι το, η παγκόσμια διαφορά εισοδήματων είναι ο κυριότερος λόγος της εμφάνισης φτώχεια, της ε, παγκόσμιας ασφάλειας και τη κυριότερη αιτία μετανάστευση. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν, χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα τις προτεραιότητε της Αυστριακής Προεδρίας και να ανταλλάξουμε απόψεις. Η Προεδρία μας λοιπόν θα κάνει ό,τι μπορεί για να δρομολογήσει τις εξελίξεις σε πολλούς ε, σημαντικούς φακέλους με λύσεις αποδεκτές για όλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας ε, στην αναπτυξιακή συνεργασία και πρέπει να δυναμώσει τη φωνή της. Οι προσπάθειες στην ε, ανθρωπιστική βοήθεια από τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε και μέλη της Επιτροπής και να ευχαριστήσω τη Βουλγαρική Προεδρία για τη δουλειά που έχει κάνει το προηγούμενο εξάμεινο. Προσπαθούμε να χτίσουμε πάνω σε τα επιτεύγματα της Βουλγαρικής και Εστονικής Προεδρίας. Η Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανθρωπιστική Βοήθεια συνεχίζει να ε, ορίζει το έργο μας για το εξάμεινο που έρχεται. Ε, η χρηματοδότηση για την ε, ανθρωπιστική βοήθεια το 2018 έχει αυξηθεί κατά 25 δισεκατομμύρια δολάρια και δεδομένων όλων αυτών θα παρακολουθούμε όλες, ε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, τις αναδυόμενες, τις παρατεταμένες και τις μακροχρόνιες ανθρωπιστικές κρίσεις. Πολλοί μιλούν για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που έρχεται. Κύριε Πρόεδρε, εσείς ξέρω πως μόλις γυρίστε από αποστολή στο νότιο Σουδάν. Ε, νομίζω πως ε, αν ε, σκεφτεί κανείς το Κονγκό και το τι γίνεται, τα εκατομμύρια θυμάτων εκεί, ε, νομίζω πως δεν θα μιλάμε για τον πόλεμο που έρχεται, αλλά για τον πόλεμο που έχει έρθει, που είναι πλέον εδώ. Υπάρχουν ορισμένες ε, ξεχασμένες συγκρούσεις, όπως έχετε πει κι εσείς και πρέπει να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που παρέχουμε, τον, την αποτελεσματικότητα του συντονισμού. Αυτό φαντάζομαι είναι αυτονόητο. Τα διάφορα μέτρα στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών αλληλοσυμπληρώνονται. Και προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια, χρειάζεται αυτό που ζητούν οι περισσότεροι οργανισμοί. Χρειάζεται δηλαδή μεγαλύτερη προσοχή ε, στην ε, επισητιστική βοήθεια. Η περσινή κρίση στην Ιεμένη, στην Σομαλία, τον Νότιο Σουδάν και την Ιγυρία θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν είχαμε δώσει τη δέουσα προσοχή σε αυτόν τον τομέα. Θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει καταστάσεις. Ε, όμως, βέβαια, οι κρίσεις αυτές ε, διονίζονται ή είμαστε μετέωροι. Αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και την αναπτυξιακή συνεργασία στο σύνολό τη. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτιέρες, δήλωσε πρόσφατα ότι πρέπει να καταρρύψουμε τους φραγμούς που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανάμεσα στην ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να ε, πασχίσουμε για βελτίωση της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας στις έξι νευραλγικές ε, χώρες, Σουδάν, Ιγυρία, Τσάτ μεταξύ άλλων. Χρειάζεται να ε, δημιουργήσουμε ένα πλέγμα συνεργασίας ανάμεσα σε αυτές τις ε, χώρες. Και πρέπει επίσης να δημιουργηθεί η σύνδεση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής βοήθειας. Περίπου το ίμιση των 65 ε, εκατομμυρίων ε, ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια είναι εσωτερικά ε, εκτοπισμένοι, εξαναγκαστικά, χωρίς τη θέλησή τους. Η 20η επέτειος των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τους εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους θα πρέπει να αποτελέσει αφετηρία για την βελτίωση των προσπαθειών από μέρους μας. Αυτά θα τα συζητήσουμε στις ε, ερωτήσει και απαντήσεις. Να πω όμως, επιτρέψτε μου, εδώ σε αυτό το σημείο, ότι η αναπτυξιακή συνεργασία έχει περιθωριοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Προς όφελος των ε, επιχειρήσεων ανθρωπιστικής ε, παρέμβασης που λαμβάνουν περισσότερη δημοσιότητα. Πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να δείξουμε τι συμβαίνει στα παρασκήνια, πίσω από τις κάμερες. Ε, το πρόβλημα, ε, η λύση μάλλον στο πρόβλημα δεν είναι η βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, είναι η μακροπρόθεσμη βοήθεια. Και επιτρέψτε μου εδώ να επανέλθω σε κάτι γενικότερο, πιο θεωρητικό, το οποίο όμως έχει αντίκτυπο στην ε, καθημερινότητα της ε, αναπτυξιακής βοήθειας έχουμε να κάνουμε με το Διεθνές Ανθρωπιστικό ε, Δίκαιο. Προσπαθούσα στην στα διαδρομία μου πριν την πολιτική να ευαισθητοποιήσω και να ενημερώσω πάνω στο ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο, στις διάφορες διατάξεις, έτσι ώστε να ε, βελτιωθούν οι συνθήκες, να υπάρχουν βασικές, ε, βασικά πρότυπα για όλους, από τον φυλακισμένο το, μέχρι τον πρόσφυγα, μέχρι τον ανήλικο. Στόχος είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες και να ενισχύσουμε ε, τον σεβασμό προς το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο. Είμαστε στον 20ο αιώνα, οπότε είναι απίστευτο το γεγονός ότι οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου όχι μόνο αυξάνονται, αλλά προσπαθούν να ε, καταργήσουν το διεθνές δίκαιο με τη μορφή ενόπλων συγκρούσεων. Πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν τη συμμόρφωση προς το ε, ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό έχουν δυσκολία πρόσβασης, δεν μπορούν να ε, πάνε σε νοσοκομεία, να ε, παράσκουν βοήθεια, περνάνε μέσα από πεδία μάχης. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και να σταθώ εδώ πολύ σύντομα στην ε, πρόσφατη συνάντησή μου με εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού στη Γενέβη πριν από δύο εβδομάδες. Η υπηρεσία αυτή λοιπόν έχει διεξάγει μελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτό που είδα με τα μάτια μου ως ε, εκπαιδευτικό πριν από χρόνια. Ότι έχει μειωθεί η ευαισθησία μας απέναντι στα βασανιστήρια. Αυτό ε, είναι απαράδεκτο. Μου λένε πως ε, τι να κάνουμε πολλές φορές είναι αναγκαίο. Και οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού μου έδειξαν τα βρήματά τους τα οποία είναι συγκλονιστικά. Πριν από 14 ή 15 χρόνια η αντίδραση ε, του κόσμου στα βασανιστήρια ήταν πολύ πιο έντονη. Ε, οι πολίτες στις χώρες όπου υπάρχουν συγκρούσεις, στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, ε, είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα βασανιστήρια, έχουν πιο έντονες αντιδράσεις, ε, δεν είναι αδιάφοροι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Μιλάμε για βασικά πρότυπα διαβίωσης τα οποία έχουμε ε, ψηφίσει το 1949 με το Σύμφωνο της Γενέβης. Πριν συζητήθηκε το θέμα αυτό πριν καν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν δεν υπήρχε ε, καν η έννοια του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Παραβιάσεις ε, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου λοιπόν τα το αντικείμενο των συζητήσεών μα με τον Ερυθρό Σταυρό και προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε ε, τους ε, διεθνεί εφορεί έτσι ώστε να να αλλάξει η κατάσταση, να ενισχυθούν οι δομές ανθρωπιστικής βοήθειας, οι δομές στήριξης τη στήριξη του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να στηρίξουμε την διεθνή ποινική δικαιοσύνη. Πρέπει να επαναλάβουμε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσει το διεθνές δίκαιο και να ε, αποδώσει ευθύνες. Το θέμα αυτό για μένα είναι η κυριότερη προτεραιότητά μου ε, και αναφέρομαι στην σεξουαλική και έμφυλη βία. Έχουμε δει ότι τον τον 20ο αιώνα οι πόλεμοι που έγιναν στην Ευρώπη αλλά και οι τελευταίοι πόλεμοι στη Γεκοσλαβία είχαν έντονα έμφυλη διάσταση. Χρησιμοποιήθηκε αυτό προς όφελος ε, των ε, αντίπαλων πλευρών. Οι γυναίκες και τα κορίτσια έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης, ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το ανθρωπιστικό μας έργο θα τηρεί υψηλές ηθικές αξίες και αρχές. Και δεν μιλώ μόνο για τη στρατολόγηση, την πρόσληψη ε, ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται υπό πολύ μεγάλη πίεση στα επιτόπου. Μιλώ για την προσωπική ηθική και την αναζήτηση των κατάλληλων ανθρώπων για αυτά τα τόσο δύσκολα καθήκοντα. Οι εκθέσεις ε, για την σεξουαλική παρενόχληση ή την κατάχρηση εξουσιών εκ μέρους των ανθρώπων που δίνουν την ανθρωπιστική βοήθεια επί τόπου ε, μας έχει εκπλήξει. Οι δωρητές ε, θα πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε να εφαρμοστούν πολιτικές μηδενικής ανοχής. Ο Κόφι Ανάν το είχε αναφέρει αυτό στην αρχή της δεκαετίας του 90 και ο Αντώνιο Γκουτέρες το αναφέρει επίσης σήμερα στην εκστρατεία του. Κάτι που μας υπενθυμίζει ότι ακόμα δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας. Η πρωτοβουλίε της διεθνούς κοινότητα για να εκριζωθεί το φαινόμενο αυτό είναι πολύ θετικέ. Ο Οργανισμό των Εθνών όμως ε, οθεί όλα τα κράτη-μέλη να αναλάβουν και τι δικέ του δράσει. Θα μπω σε περισσότερε λεπτομέρειε σε ό,τι αφορά το φύλλο αργότερα. Όλη μα η εξωτερική, η ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να έχει τι γυναίκε στο μυαλό τη στο επικέντρό τη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα αναπαραγωγική υγεία. Να αναφερθώ και στα διμερεί προγράμματα τα οποία έχουμε στήσει για να αντιμετωπίσουμε ε, το φαινόμενο του ακροτηρισμού γενετικών οργάνων κοριτσιών. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μας τυχιώνει εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε προσπαθήσει να το εντοπίσουμε και να το αναδείξουμε. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Κατάργηση των Διακρίσεων Αντίον των Γυναικών έχουμε αναλάβει να εξασφαλίσουμε ίσα δικαιώματα και να επιτρέψουμε στις γυναίκες να αποφασίζουν αυτόνομα για το πόσα παιδιά θα έχουν, πότε θα τα αποκτήσουν και να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Η Επιτροπή επίσης αναφέρει ότι τα δικαιώματα των γυναικών στην εκπαίδευση μέσω πρόσβαση σε ιδιαίτερη ε, στοχευμένη πληροφόρηση συμπεριλαμβανομένη και πληροφόρηση και συμβουλών για οικογενειακό προγραμματισμό είναι απολύτω απαραίτητο. Οι δημογραφικέ εξελίξει καθιστούν απαραίτητη αυτή την προσέγγιση και η εκπαίδευση των γυναικών, καθώς επίσης και η ανάπτυξη του βιωτικού επίπεδου, είναι απόλυτα σημαντικά στοιχεία προκειμένου να μειωθούν οι δημογραφικές πιέσεις. Τώρα, θα αναφερθώ στο θέμα του, ε, της, της κατάστασης μετά το, κοστό, μετά το κοτόνο. Στις 22 Ιουνίου το Συμβούλιο αποφάσισε να ε, συμφωνήσει μια, σε μια κοινή διαπραγματευτική εντολή για να ξεκινήσουν ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διαπραγμάτευση μια νέα συμφωνία με τι χώρε ΑΚΕ ω μια βάση για τι μελλοντικέ σχέσει μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των 79 χωρών ΑΚΕ. Στόχο είναι μια ε, ισότιμη εταιρική σχέση σφαιρική που θα λαμβάνει υπόψη τη νέα κατάσταση, τι νέε προκλήσει με στόχο τη μείωση τη φτώχεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο ιδιωτικό τομέα και η κοινωνία των πολιτών θα είναι σημαντικοί παίκτε προκειμένου να δημιουργηθούν θέσει εργασία και να βελτιωθεί η διακυβέρνηση σε αυτό το καινούριο πλαίσιο συνεργασία. Η προτινόμενη εντολή ε, προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε ένα, στα θεμέλια τα οποία είναι κοινέ αξίε και στόχοι, όπω για παράδειγμα η αποτελεσματική εφαρμογή της Ατζέντα ε, ε, 2030 για την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Τώρα, να αναφερθώ σε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό, το πολιτε δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 για τις ερωταπαντήσεις να σας πω ότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι δική μου αρμοδιότητα, αρμοδιότητα του δικού μου Υπουργείου Παρ' όλα αυτά πρέπει να το σχολιάσω. Με σημαντικές αλλαγές στην ε, διάρθρωση της, ε, της Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η Πολλά κράτη-μέλη ζητούν να αντιμετωπίσουμε το ευρωπαϊκά την μετανάστευση, οπότε η Κομισιόν προτείνει να μειώσουμε σημαντικά τον αριθμό των οργάνων εξωτερικής χρηματοδότησης. Το νέο χρηματοδοτικό όργανο που θα ονομάζεται NDICI, ε, Γειτονία, Ανάπτυξη και διεθνή συνεργασία, ε, θα περιλαμβάνει θεματικά και γεωγραφικά μέσα το βασικό μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω εγώ είναι ότι ε, οι στόχοι βιώσιμη ανάπτυξη δεν έχουν μόνο εξωτερική διάσταση αλλά και εσωτερική διάσταση. Η πεπατημένη δεν είναι ε, πλέον λύση. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τους λαούς και τις κυβερνήσεις. Πρόσφαση στα, να δείτε πρόσβαση στα, βήματα, στα θύματα, η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα είναι αρκετές για να αντιμετωπίσουμε τα δράματα τα οποία εμφανίζονται. Να σας πω τα λόγια κάποιου που ακόμα έχει πολλά πράγματα να μας πει. Θα μπορούσε να γιορτάζει τα 100 χρόνια της ζωής του σήμερα, ε, αλλά έχασε, ε, δεν είναι πια ζωντανός μαζί μας, ο Νέλσον Μαντέλα, Είχε πει ο Νέλσον Μαντέλα, που είναι ένας άνθρωπος που ακόμα μας εμπνέει, ε, για το κουράγιο και την επιμονή. Ε, ήταν εκπληκτικής υπομονής και επιμονής άνθρωπος και υπό τρομακτική πίεση δεν έσπασε ποτέ. Είχε πει το εξής. Ε, όπως το απαρχάει και η λουδία έτσι και, και, η δουλεία έτσι και η φτώχεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Ε, είναι ανθρώπινη προέλευσης και μπορεί να εκριζωθεί με πράξεις ανθρώπων. Η εκρίζωση της ε, φτώχειας είναι και θα είναι ο πιο σημαντικός στόχος των κοινών μας προσπαθειών σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Υπουργέ όσον αφορά το τελευταίο για την μείωση της φτώχειας και τη σχέση με την αναπτυξιακή ε, πολιτική. Εμείς ε, εδώ πάντα το λέμε, συμφωνούν όλες οι ομάδες και κάνουμε ό,τι μπορούμε με τον ρόλο που έχουμε, που είναι νομοθετικός όπως είπατε και εσείς ότι μέσα διαθέτουμε, προσπαθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για την μείωση της φτώχειας. Ε, υπάρχει το όνομά σας στον κατάλογο ομιλητών. Ε, αλλά να συνεχίσω με ένα σχόλιο. Είπατε διάφορα πράγματα πάνω στα οποία έχουμε δουλέψει κι εμείς πολύ. τον Nexus. Το βασικό θα είναι η χρηματοδότησή του στο μέλλον. Γιατί είναι δύσκολο να χρηματοδοτούμε προγράμματα χωρίς πόρους. Στην Ουγκάντα, για παράδειγμα, ε, που ασχολούνται με πάρα πολλούς πρόσφυγες, γυναίκες και παιδιά από το Σουδάν. Όπως είπατε, έχουμε μια κρίση, βάζουμε πάρα πολλά χρήματα, μετά λέμε χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα και όλα γίνονται έτσι βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή δεν καταφέρουμε να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα ή να δεσμευτούμε μακροπρόθεσμα. Αυτά που είπατε για τα βασανιστήρια επίση είναι θλιβερό, έτσι. Η ιδέα ότι οι νέοι που σπουδάζουν διεθνείς σχέσεις στις χώρες μας είναι λιγότερο ευαισθητοποιημένοι σήμερα στα θέματα των ε, βασανιστήριων είναι πολύ θλιβερό, πράγματι. Ίσως γιατί τα τελευταία 20 χρόνια αρχίσαμε να θεωρούμε κανονικότητα την ε, συμπεριφορά αυτή. Και η χώρα μου φυσικά είναι υπεύθυνη για αυτό που έγινε με τους κρατούμενους που μυστικά ε, πήγαιναν σε άλλες χώρες για βασανιστήρια. Μετά το 1945 ακριβώς επειδή έγιναν αυτά που έγιναν όλοι δημιουργήσαμε το δίκαιο για να μην ξαναγίνουν. Έπειτα η σεξουαλική βία που αναφέρατε επίσης είναι φοβερό και έχουμε βραβείο εμείς για την ελευθερία σκέψης και τα ανθρώπινα δικαιώματα και πριν από λίγα χρόνια απενεμήθη στον ε, δόκτωρο Μακβέγγε ο οποίος είναι από το Κονγκό και ο οποίος ε, φροντίζει ε, ως γιατρός να βοηθήσει οι γυναίκες και κορίτσια θύματα τέτοιας ε, σεξουαλικής βίας, βιασμών. Το κάνει λοιπόν και τον βραβεύσαμε. Βραβεύσαμε και δύο γυναίκες οι οποίες και αυτές ήταν θύματα στο Ιράκ βιασμών. και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της ατιμορρησίας. Όταν υπάρχει η ειρήνη και πάλι, όταν η Ντάες φτάσει στη δικαιοσύνη, μετά τι θα κάνουμε αυτό έχει μεγάλη σημασία επίσης. Αλλά σίγουρα και άλλα ζητήματα θα θέλουν να θίξουν οι συνάδελφοι. Θα αρχίσουμε από τον κύριο Νόιζορ, ο οποίος καθιστά τον ε, κύριο Γκερέρο δεν μπορεί να είναι εδώ εκείνο. Νομίζω ότι μιλάει σε μια ομάδα νέων για τα ζητήματα ανθρωπιστική βοήθειας. Πολύ σημαντικό μετά από τόσα μα είπατε, η συνειδητοποίηση αυτή των νέων έχει σημασία. Οπότε ο κύριος Νόιζερ θα μιλήσει εκ μέρου του, μετά ο κύριο Πόλο Ρούμπεκ και μετά οι υπόλοιποι. Παρακαλώ. Ναι, θα μιλήσω γερμανικά. αν και υπάρχουν διαφορές στην κοινή μας γλώσσα ανάμεσα σε εμά και σε εσά. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Μιλώ εκ μέρους του Ενρίκη Γκερέρο Σαλόμου, ο οποίος ε, δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι εδώ. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ να σας ακούσει, είμαι σίγουρος. Ο κύριο Σαλόμ και εγώ συμφωνούμε και έχουμε σύμφωνα απόψεων. Νομίζω πως η παρουσίασή σας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτά που λέτε. Η καταπολέμηση της ε, ακραίας φτώχειας είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να ανήκει στους αναπτυξιακούς στόχους ε, στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, ε, πρέπει να ομολογήσω ότι το βάρος που έχει δοθεί σε κάθε μία από τις προτεραιότητες ε, με βρίσκει ε, δεν με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Το βάρος που έχει δώσει η Αυστριακή Προεδρία στην ε, μετανάστευση προ την Ευρώπη ε, είναι για μας λίγο υπερβολικό. Είπατε επίση πως έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλές προκλήσεις, μακροπρόθεσμες προκλήσεις. Θεωρώ πως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς διότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις είναι τεταμένες, ε, υπάρχουν έντονες διαφωνίες και νομίζω πως μας λείπει ένα πλαίσιο. Μας ε, αναφέρεται επίσης για το πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε μετά το κοτονού. Και αυτό μπορώ να το προσυπογράψω. Χρειάζεται καλύτερο συντονισμό στις ευρωπαϊκές μας θέσεις. Ε, πολύ ωραίο όλο αυτό, όμως θα ήθελα να κάνουμε περισσότερα, να είμαστε πιο δυναμικοί. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε πεπισμένοι ότι η συμφωνία του κοτονού ήταν ε, επιτυχής. Χρειάζεται ε, όμως ε, να γίνουν περισσότερα, να υπάρχει καλύτερη διακυβέρνηση, μεγαλύτερη συμμετοχή των ε, κοινοβουλίων, καλύτερη συνεργασία με τις χώρες ε, ΑΚΕ. Αυτό πρέπει να ε, μην το θεωρούμε δεδομένο ότι έχει ολοκληρωθεί με τη Συμφωνία του Κοτονού. Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Ήμουν συντάκτης της σχετικής έκθεσης και πρέπει να σας πω ότι αν η Ρωσία, οι Ηνωμένες η Κίνα ε, είχαν υπογράψει μια τέτοια σύμβαση με 79 χώρες, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά, θα τα είχαν αλλάξει όλα. Ε, η χρονική αυτή στιγμή είναι μια εποχή δύσκολη. Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και την Κίνα είναι επίσης δύσκολες. Δυσκολευόμαστε να βρούμε μια κοινή θέση εδώ μεταξύ μας. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να δώσουμε τη δέωσα σημασία συμφωνία του Κοτονού και να την προχωρήσουμε αν θέλουμε να καταφέρουμε οτιδήποτε. Τώρα νομίζω πως ε, θίξατε επίσης πολύ σημαντικά θέματα. Πρέπει να διαπραγματευτούμε με τις ίδιες τις χώρες ε, κατευθείαν. Πρέπει να δώσουμε όμως ευρωπαϊκή λύση και όχι ο καθένας να κάνει αυτό που νομίζει. Ευρωπαϊκή λύση λοιπόν ε, στα προβλήματα και έχουμε θετικές ενδείξεις, θετικά μηνύματα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στην ε, στρατηγική μας. Αυτή τη στιγμή στην Αιθιοπία λαμβάνουν χώρα δραματικές πολιτικές εξελίξεις ε, και στην Ερυθρέα επίσης και είναι πιστεύω μια τεράστια ευκαιρία την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Ε, πολύ απλά θα σας τα πω. Η μετανάστευση από την Αιθιοπία και την Ερυθρέα θα μπορούσε να μειωθεί αν οι λόγοι για τους οποίους λαμβάνει η χώρα αυτή η μετανάστευση ε, εξαφανιστούν, αν δεν γίνονται πολιτικές διώξεις. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν ε, όμως ε, σας παρακαλώ να μας ε, στηρίξετε. Η Αυστριακή Προεδρία πρέπει να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Um, um, ευχαριστώ πολύ. Ο Πόλο Ρουμπίκ. Σας ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας καλωσορίζουμε σήμερα, κυρία Υπουργέ, διότι ε, η αναπτυξιακή πολιτική και η αναπτυξιακή συνεργασία είναι ε, όρια αλληλένδετη. Πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να ε, στεφθούν οι προσπάθειές μας με επιτυχία και να επιτύχουμε τους στόχους μας. Έχουμε συζητήσει εκτενέστατα τον προϋπολογισμό του 2019 οι συνάδελφοί μου και εγώ. Ο συνάδελφος Άρνε Λίτς έχει συντάξει μια εξαιρετική έκθεση, δίνει έμφαση στην ε, βοήθεια για υγεία, για εκπαίδευση, για κατάρτιση, για το περιβάλλον, ε, για τη διάσταση του φίλου, για την ισότητα. Είναι όλα αυτά στόχοι τους οποίους θα επιτύχουμε μέσω της αναπτυξιακής συνεργασίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Ε, πρέπει να φροντίσουμε για τον ε, επισητισμό, το σωστό επισητισμό και εδώ πρέπει να κάνουμε πολλά. Νομίζω πως ε, πρέπει η διατροφή να, είναι, ε, να μπει στις προτεραιότητες μας. Ο στόχος νούμερο 6 επίσης πρέπει να ε, ανέβει σε, ως προτεραιότητα. Η βελτίωση των υγειονομικών συνθήκων στα νοσοκομεία είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Αυτή τη στιγμή δεν γίνονται πολλά και νομίζω πως έχουμε μάθει από την πολιτική συνοχής εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης πως ε, υπάρχει ανάγκη να δώσουμε έμφαση στην ύπεθρο σε λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες και να δώσουμε τη δυνατότητα ε, σε μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ε, δημόσιους ανοιχτούς διαγωνισμούς. Χρειάζεται να βελτιωθεί λοιπόν η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η πρόσβαση των ίδιων των πολιτών σε δυνατότητες χρηματοδότησης και στήριξης. Αυτή την πολιτική θα μπορούσαμε να την προσαρμόσουμε και να την εφαρμόσουμε στις ε, χώρες της Αφρικής και όλες τις χώρες ε, στις οποίες δραστηριοποιούμαστε ε, με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ε, το 2019 στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, όμως ελπίζω με το νέο πρόγραμμα πλαίσιο της Αυστριακής Προεδρίας να προχωρήσουμε. Ελπίζω η δική σας Προεδρία να ε, το προχωρήσει. Αυτά από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθετε. Thank you. Ευχαριστούμε, ο Σάρλ Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω την ε, Προεδρεύουσα του Συμβουλίου που θέτεται ζητήματα που μας απασχολούν μεταξύ άλλων οι σε βάρος των γιακών. Θέλω να θυμίσω ότι την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο υιοθετήσαμε μια έκθεση για τους γάμους που γίνονται κατανακαστικά σε πολύ νερή και των κοριτσιών. Από ό,τι φαίνεται 50 εκατομμύρια νέων κοριτσιών και αγόρια, αλλά κυρίως βέβαια γυναίκες, υφίσταται αυτή τη μάστιγα. Δεν είναι λίγο πράγμα και είναι κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά γνωστό και έχει να κάνει και με τις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς έχουμε επιμείνει ότι πρέπει να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε εμείς ίδιοι να αποκτήσουμε τους κατάλληλου κανόνες γιατί δεν έχουν στην ομοθεσία τους όλες οι χώρες τον περιορισμό των 18 ετών, δηλαδή να μην υποχρεώνεται να παντρευτεί κανένα κορίτσι κάτω των 18. Ενώ αυτό είναι το πρότυπο που είναι αποδεκτό παγκοσμίω. Και τελικά ε, προσφεύγουμε στον ΟΗΕ, στην UNICEF και άλλες οργανώσεις του ΟΗΕ για να βοηθήσουν. Και το ίδιο μπορούμε να πούμε και για την κλιτερδεκτομή που γίνεται στα κορίτσια. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας κι εσείς ότι είναι απαραίτητο να καταπολεμηθεί αυτή η μάστιγα και να δώσετε στρατηγική προτεραιότητα. Κάτι άλλο τώρα. Αναφερθήκατε στη διάκριση των εξουσιών και αναφερθήκατε στο Μοντεσκέ. Εγώ είπα, «Ε, αυτό είναι για μας ε, μελωδία στα αυτιά μας. Ε, όντως, εμείς είμαστε περισσότερο σε θέση να το κρίνουμε, γιατί και εμείς ταλαιπωρούμαστε από αυτή τη σχέση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το πρόβλημα όμως που έχουμε δεν είναι τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι περισσότερο με τις χώρες μέλη. Γιατί οι χώρες μέλη συμφώνησαν να γράψουν στην Ευρωπαϊκή Συνένεση για την Ανάπτυξη συγκεκριμένες δεσμεύσεις σημαντικές και φιλόδοξες. Όταν όμως καλούμε τις χώρες μέλη να μας δείξουν τι έχουν κάνει πώς έχουν υλοποιήσει τους στόχους αυτούς για τους οποίους δεσμεύτηκαν, εκεί ξαφνικά κανένας δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Οπότε, κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας, θα ήθελα, παρακαλώ, να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος, ορίζοντας τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου στον έλεγχο, κυρίως για ό,τι έχει να κάνει με τις επιμερισμένες ευθύνες και αρμοδιότητες. Γιατί έχουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συμπεριλαμβάνει και αυτή τη διάσταση. Όμως, για να είμαστε συνεπείς και για να υπάρχει και συνοχή σε αυτά που κάνουμε, θα πρέπει όλοι να βάλουν ο καθένας το δικό του πετραδάκι. Οπότε και οι χώρες μέλη θα έπρεπε να έρχονται εδώ στην Επιτροπή μας και να εξηγούν με ποιο τρόπο ε, σκοπεύουν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει. Εδώ και 40 χρόνια λέμε παραμύθια για το περίφημο 0,7%. Οι χώρες το έχουν βάλει στην νομοθεσία του, στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, άλλες δεν τα καταφέρνουν, γιατί δεν υπάρχει σωστή μέθοδος. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά. Και για το πολιτές ε, ε, δημοσιονομικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε το ρόλο το συντονιστικό στο νομοθετικό έργο. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα για το πώς βλέπετε εσείς την μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το Συμβούλιο. Πώς βλέπετε τις συνομιλίες με τους συναδέρφους σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και κυρίως με το μηχανισμό των ενιαίων χρηματοδότησης. Βλέπετε να μπαίνουμε σε τριμερή διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα αποτελέσει αυτό μια πραγματική προπτική επίλυση των ζητημάτων, γιατί δεν τον αποφύγουμε τον τριμερή διάλογο. Πρόεδρος. Πώς έχω ακόμα στον καταλογό μου άλλους δύο. Να ακούσουμε και τις άλλες δύο ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε. Θα έχετε απλό το χρόνο για να απαντήσετε σε όλα. Ξέρω, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Η Μαρία Χόιμπουκ πρώτα. Παρακαλώ. Θα σας τα θυμίσουμε τα έχετε ξεχάσει τις ερωτήσεις δηλαδή. Μαρία. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κυρία Υπουργέ. Η παρουσίασή σας ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Άκουσα πολλά τα οποία προσυπογράφω ίδια και νομίζω πως ε, πραγματικά χρειάζεται στήριξη και συνεργασία αν θέλουμε η ανθρωπιστική βοήθεια να έχει αποτελέσματα. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στην αναπτυξιακή και στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά πρέπει να ανοίξει και μια δημόσια διαβούλευση πάνω σε αυτό το θέμα. Διάβασα με προσοχή το πρόγραμμα της Αυστριακής Προεδρίας και το πρώτο που μου έκανε εντύπωση είναι η πρώτη παράγραφος του κεφαλαίου για την ανάπτυξη, όπου λέει ε, σχεδόν κατά λέξη ότι ως αντίδραση στο μεταναστευτικό ζήτημα η σύνδεση ανθρωπιστικής βοήθειας με μακροπρόθεσμης ε, αναπτυξιακής βοήθειας και αναπτυξιακών... μέτρων θα δημιουργήσει προοπτικές για νέες ε, συνέργειες. Η Αυστρία ε, θα κάνει ό,τι μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση και θα φροντίσει για τη σύνδεση ε, της επικοινωνίας ανάμεσα σε τρίτες ε, χώρες και την επαναπροώθηση ατόμων σε αυτές τις χώρες. Αυτά σχεδόν κατά λέξη, δηλαδή συνδέεται την αναπτυξιακή συνεργασία με το μεταναστευτικό ζήτημα. Και τώρα μας είπατε ότι προσπαθήσατε ε, πριν μπείτε στην πολιτική να μεταδώσετε ως εκπαιδευτικό σε βασικές ε, έννοιες για βασικά ε, βασικά πρότυπα. Αυτά είναι μεταξύ άλλων η ουδετερότητα και η επιχειρησιακή ανεξαρτησία. Και με αυτή την πρόταση όμως ε, στο, στο σχέδιο της Αυστριακής Προεδρίας τα πατάτε όλα στα σκουπίδια. Από ό,τι καταλαβαίνω εγώ βλέπω ότι τα κυρώνετε όλα αυτά που λέτε πως πρεσβεύετε. Δεν μπορώ να το πιστέψω σχεδόν. Δεύτερον, εάν η μετανάστευση είναι τόσο ε, μπροστά στη λίστα των προτεραιοτήτων σας, ε, τότε, μια που αναφέρετε και τη Συμφωνία του Κοτονού, ε, μου φαίνεται λίγο δύσκολο να καταλάβω τι ακριβώς εννοείται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέχεια ε, πετάμε τον μπαλάκι στη μετανάστευση και το συνδέουμε με όλες τις υπόλοιπες πτυχές της πολιτικής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εσείς πώς θα καταφέρετε να ε, διασφαλίσετε αυτήν την ισορροπία όταν αποτελείτε μέλος ε, μιας κυβέρνησης ε, στην Αυστρία όπως όλοι την γνωρίζουμε. Κατά την προεκλογική εκστρατεία σας Ο καγκελάριος Κούρτς μίλησε εκτενέστατα για αύξηση των κονδυλίων για ε, βοήθεια επιτόπου. Και τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε ήταν έτσι ωραιοποιημένα θα έλεγα. Ήταν κάποια ε, γραφήματα με τους ε, δωρητές, όμως ήταν κάπως έτσι φτιαγμένα, ρετουσαρισμένα, έτσι ώστε να φαίνεται η Αυστρία ανάμεσα στους μεγαλύτερους δωρητές ανθρωπιστικής βοήθειας. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, τα πιστεύετε οι ίδιοι αυτά. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω, την, ε, για την, ε, να πιστέψω τις στατιστικές αυτές όταν έχουν τόσο ρετουσαριστεί. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που ο καγκελάριος ο ίδιος ε, παρουσιάζει αυτές τις πληροφορίες έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλος η Χέντι Χάουταλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ στην Επιτροπή μας. Σημείωσα πόσο καλά γνωρίζετε τα θέματα της διεθνούς ανθρωπιστικής ε, βοήθειας που τα κατέχετε καλά και πόσο πολύ σας ενδιαφέρουν. Κάποιοι ευρωβουλευτές και εγώ ίδια απευθυνθήκαμε στην κυρία Μογκερίνη με πρόταση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει διοικό εκπρόσωπο για θέματα ανθρωπιστικού δικαίου και ίσως και για την ποινική δικαιοσύνη που αναφέρατε. Ίσως να μην είναι ο μόνος τρόπος για να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση και στήριξη στο, ε, στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, αλλά θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για τη δικιά σας τη γνώμη. Δηλαδή, εσείς ε, τι πιστεύετε, τι μηχανισμούς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με αυτά. Για τα βασανιστήρια τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να είναι πάνω πάνω στην ημερήσια διάταξη. Και χαίρομαι που το είπατε. Έρχομαι τώρα στο θέμα της μετανάστευσης. Κοίταξα στη Wikipedia τη σελίδα σας και είδα ότι το Σεπτέμβριο του 2015 με τη λεγόμενη μεταναστευτική κρίση εσείς αναφερθήκατε σε νέους Άραβες οι οποίοι δεν καταφέρουν να βρουν γυναίκα, σύζυγο, ότι δεν μπορούν να κρατήσουν το ρόλο τους στον παραδοσιακό στις κοινωνίες τους και μιλήσατε για τον έλεγχο της τεστοστερόνη κλπ. Εντάξει, μπορείτε να έχετε αυτή την άποψη, αλλά εγώ επειδή εκπροσωπείτε την Προεδρία, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, τι λύσεις βλέπετε εσεί. Αυτά όπως τα εκφράσατε, δεν νομίζετε ότι δεν διέπονται από αρκετή αντικειμενικότητα. Ωραία, αυτές ήταν οι ερωτήσεις των συναδέρφων. Παρακαλώ. <coughs> Αγαπητέ κύριε Νόιζερ, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, στήριξη που δείχνετε στο πρόγραμμα της Προεδρίας μας και θα ήθελα να αρχίσω απαντώντας την ερώτησή σας σχετικά με, να το βρω μισό λεπτό, με την περίοδο μετά τον Κοτονού, τη Συμφωνία του Κοτονού. Η συμφωνία που διαπραγματευτήκαμε είχε έναν ε, κατάλογο με ανθρωπιστικά κριτήρια, εργασιακά κριτήρια και άλλα και αποδείχθηκε η αξία του. Ε, οδήγησε σε ε, θετικές εξελίξεις και αποφασιστική σημασία είναι ότι θέλουμε να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να πάμε ακόμα παραπέρα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση ευρωπαϊκή για την επιστροφή, πανεσδοχή των προσφύγων. Εσείς ε, μιλήσατε για ε, διμερείς λύσεις, όμως το καλοκαίρι του 2015 έγινε πολλής λόγος για ε, την ευρωπαϊκή λύση. Βρέθηκε μια ευρωπαϊκή λύση και βλέπουμε τώρα ότι τρία χρόνια αργότερα η τάση είναι να επιστρέφουμε στις διμερείς συμφωνίες. Να σας παραθέσω και τα λόγια της καγκελαρίου Μέρκελ πάνω σε αυτό, ότι η ευρωπαϊκή λύση πρέπει, κατά την άποψή μας, ε, να αφορά το ότι πρέπει να αντιληφθούμε πως ε, τα μέσα που έχουμε αναπτύξει για να αντιμετωπίσουμε μεταναστευτικά ζητήματα ε, είναι λύσεις οι οποίες ε, δεν λαμβάνουν υπόψη την παγκοσμιοποίηση. Είναι λύσεις της δεκαετίας του 80 παροχημένες. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουν τα δεδομένα, να επικαιροποιήσουμε την πολιτική μας, διότι δεν είναι πλέον επίκαιρη. 65 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους, υπάρχουν τεράστια ποσοστά ανεργίας, υπάρχουν τρόμερα προβλήματα και στην εκπαίδευση, φτώχεια. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να δώσουμε έμφαση στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση λύνει τα πάντα. Ε, όμως υπάρχουν προβλήματα. Οι περισσότεροι ε, δεν βρίσκουν δουλειές παρότι έχουν ε, σπουδάσει. Έχω δει και έχω μιλήσει με πολλούς ε, φοιτητέ στη Λιβύη, στην Αίγυπτο που μετά τι σπουδέ τους δουλεύαν σε καφετέριες γιατί δεν μπορούσαν να βρουν άλλη δουλειά. Εδώ λοιπόν υπάρχει διαφορά. άλλε οι λύσεις και άλλα τα δεδομένα στην Ευρώπη και άλλα εκεί. Χρειάζεται να ε, δούμε τις διαφορές και πρέπει να συνδεθεί η εκπαίδευση και με το μεταναστευτικό. Αυτό που προσπαθούμε είναι από τη μία να θέσουμε τις βάσεις για τη δημιουργία μέσων που θα ε, φέρουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες και δεν θα, δεν θα πηγαίνουν οι πολίτες προς τις υπηρεσίες. Τα μέσα που έχουμε σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, προέρχονται από τη δεκαετία του 80 και είναι παροχημένα. Δεν ισχύουν πλέον τα ίδια δημογραφικά ε, στοιχεία. Ε, έχει αλλάξει η κατάσταση. Ε, σε πολλές ε, χώρες της Βόρειας Αφρικής βλέπουμε ότι υπάρχουν απόφοιτοι με εκπαίδευση άνεργοι. Διότι υπάρχει έλλειψη εργατικού δυναμικού και όχι έλλειψη πτυχιούχων. Όμως, σήμερα βλέπουμε πως υπάρχουν στη διάθεσή μας μέσα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις ε, ανάγκες της εποχής. Η παγκοσμιοποίηση λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη στη δημιουργία νέων μέσων αντιμετώπισης, νέων πολιτικών. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει εφεύρει τη ε, χρυσή λύση. Πρέπει όμως να γίνει και άλλη δουλειά. Να αναγνωριστεί η παγκοσμιοποίηση ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της ε, μετανάστευσης. Να δώσουμε έμφαση στην υποσαχάρη Αφρική και στην Νοτιοανατολική Ασία. Να δούμε γιατί μετακινεί το πληθυσμός. Δεν επαρκούν όμως τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα. Τώρα, ε, σας ευχαριστώ πολύ που αναφέρατε την Αιθιοπία και την Ερυθρέα. Ευτυχώς, δόξα το θα έχουν γίνει πολλά θετικά ε, τον τελευταίο καιρό και νομίζω πως βρισκόμαστε ενώπιον μιας μεγάλης αλλαγής. Ε, έχουν μειωθεί ε, τα θύματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υποσαχάρη Αφρική, να σας πω ότι έχω δουλέψει ίδια εκεί πολύ και νομίζω πως όντως κάτι κινείται. Αυτά που έχω παρατηρήσει στην Αφρική τα τελευταία χρόνια είναι ότι η περιφερειακή συνεργασία είναι κέρια σημασίας. Είναι απαραίτητη, διότι στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας λύνονται πάρα, πάρα πολλά προβλήματα. Εδώ βέβαια υπάρχουν διαφορές στην Αφρική. Βλέπουμε ότι στη Βόρεια Αφρική τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα τα αναφερθήκατε στην ε, επιστροφή των ε, προσφύγων, επανεισδοχή. Αυτό που πιστεύω πρέπει να δούμε είναι οι χώρες διέλευσης και το τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Ε, η λύση Ερντογάν είναι και αυτή μία λύση από τη δεκαετία του 80 θα έλεγα. Ε, η πολιτική αυτή είναι επίσης παροχημένη. Η Νιγηρία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κρατήσει τα μεταναστευτικά ρεύματα προς ε, την Ευρώπη. Όμως πρέπει να αλλάξει και η πολιτική μας. Ε, δεν είναι η κατάσταση ίδια με αυτή πριν από 20 χρόνια. Υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και σίγουρα το καλοκαίρι του 2015 ήταν, ε, το, ήταν η αφετηρία για αλλαγή πλεύσης. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν για να φύγουν, για να έρθουν στην Ευρώπη. Και εδώ να επαναλάβω. Ο κόσμος μένει στα χωριά του, μένει στις πατρίδες του, μένει στις γειτονιές του, στην πόλη του, εάν υπάρχει εγγύηση για ελάχιστες, ελάχιστες παροχές ε, ρεύματος, ε, νερού, υγείας, εκπαίδευσης. Αυτό το λένε όλοι, όλες οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ε, υπάρχουν μέρη όμω στην Αφρική που, έχουν ρεύμα, που δεν έχουν ρεύμα ή όπου έχουν, έχουν τρει-τέσσερι ώρε την ημέρα που δεν έχουν πόσιμο νερό. Ε, υπάρχουν προβλήματα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της Αφρικής ε, με την ηλεκτροδότηση. Εάν λοιπόν υπάρχει ένα εγγυημένο ελάχιστο παροχών, τότε θα άλλαζαν ε, τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε αυτήν την ελάχιστη βοήθεια. Επίσης, αυτό θα βοηθήσει στην καταπολέμηση της ακραίας ένδυας. Ελπίζω τώρα να απάντησα στις ερωτήσεις σας, ε, κύριε Νόιζερ. Κύριε Ρούμπιγκ, η σειρά σας για απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τα εκτιμώ πολύ. η εξωτερική πολιτική και η ε, αναπτυξιακή βοήθεια, η ανθρωπιστική βοήθεια πάνε χέρι με χέρι. Σίγουρα, δίχως άλλο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται και στο νότιο ημισφαίριο και είναι ορατά τα αποτελέσματα ε, που έχει σημειώσει για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας. Εγώ, εδώ, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να πάμε ακόμα παραπέρα. Υπάρχουν δυστυχώς ε, προβλήματα στη δομή των στη διάρθρωση την ίδια των σχέσεων ανάμεσα στις ε, χώρες που ε, είναι δωρητές και στις χώρες που είναι παραλήπτες ανθρωπιστικής βοήθειας και αυτό πρέπει να αλλάξει. Επίσης, θα ξανά ε, τονίσω το θέμα της ε, σωστής διατροφής, το επισητιστικό ζήτημα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στα δύο άκρα του φάσματος. Από τη μία υπάρχει πολύ μεγάλη παχυσαρκία και από την άλλη ποσιτισμός. Και αυτά δεν αφορούν μόνο ένα ημισφαίριο, νότιο, βόρειο, ανατολικό, δυτικό. Αυτό το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και στην Ασία επίσης. Μετά, εκπαίδευση και κατάρτιση μας είπατε πως πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι στα αποτελέσματα, στην πρακτική εκπαίδευση. Ε, έχουμε δει όμως ε, πολλές περιπτώσεις αραβικών χωρών όπου υπάρχει ανισορροπία ανάμεσα στη θεωρητική και στην πρακτική εκπαίδευση και αυτό οδηγεί σε μαζική μετανάστευση. Επίση, ίδρευση, αποχέτευση, εγκαταστάσει. Ε, θέματα ισότητας. Πρέπει να διασφαλίσουμε ελάχιστες ε, συνθήκες ε, διαβίωσης, να διασφαλιστεί προστασία ε, των γυναικών και των κοριτσιών. Να επανέλθω επίσης στο πρόβλημα ίδρευσης και αποχέτευσης, ξεχωριστών εγκαταστάσεων ίδρευσης και αποχέτευσης στις εγκαταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων. Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Ο Bill Gates με το ίδρυμά του προσπαθεί να βρει μια λύση στο πρόβλημα αυτό, το οποίο δεν αποτελεί μόνο η θέμα υγείας, αλλά και θέμα της ε, ασφάλειας ε, των ε, γυναικών. Πρέπει να υπάρχουν χωριστές τουαλέτες ανδρών και γυναικών, λοιπόν, στα, στις εγκαταστάσεις προσφύγων. Μετά, να σας υπενθυμίσω ότι τη δεκαετία του 70 ένα μεγάλο ποσοστό του χρέους ε, των ε, χωρών στο νότιο ημισφαίριο είχε προέλθει από την, κρίση, από την πατρελαϊκή κρίση. Γιατί, διότι μεταξύ άλλων είχα, είχε πέσει κατά πολύ η τιμή των πρώτων υλών και αυτό συνδέθηκε και με τη μετανάστευση. Τώρα, για να δούμε την κατάσταση στην Αφρική. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές ομάδες που προσπαθούν μέσω της Λιβύης να πάνε στην Αφρική. Άνθρωποι από την Ιγυρία, από τον Μπαγκλαντές και το Πακιστάν. Όχι από εκεί που νομίζετε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από χώρες οι οποίες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από την αλλαγή στην τιμή του πετρελαίου. Ε, τα κράτη του κόλπου είναι μεγάλος εργοδότης και είναι μάλιστα ε, ο κυριότερος, ο πρώτος στόχος από πολίτες αυτών των ε, προαναφερθέντων κρατών. Να δούμε και μία άλλη περίπτωση. Η Αγκόλα στην Αγκόλα τα τελευταία χρόνια έχουν, πάει, έχουν μεταναστεύσει περισσότεροι άνθρωποι από την Ευρώπη παρά ε, άνθρωποι από την Αγκόλα προς την Ευρώπη. Και αυτό γιατί έχει, ε, η απάντηση βρίσκεται στην ενέργεια, στο πετρέλαιο. Πρόκειται για μια διαρροή εργατικού δυναμικού προς τις πλούσιες χώρες, ε, το οποίο φυσικά συνδέεται και με την ενεργειακή κρίση. Αυτά τα ξέρουμε. Υπάρχουν αρκετές μελέτες, όχι καινούριε, από την δεκαετία του 80. Και μου κα... πραγματικά θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κερδίζουν 200-300 δολάρια δουλεύοντας στις χώρες του Περσικού κόλπου, αλλά καταφέρνουν και στέλνουν τα μισά στα σπίτια τους, στην πατρίδα τους στους δικούς τους. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι με το συνάλλαγμα δηλαδή, με τα εμβάσματα μπορεί να δοθεί μια λύση στο θέμα και το πρόβλημα του χρέους. Όταν οι ξενιτεμένοι στέλνουν εμβάσματα πίσω. Μετά, να απαντήσω στις ερωτήσεις του Σαλ Αν κατάλαβα καλά αυτό που ρωτήσατε, Άιστα από την Αλσατία. Λουξεμβούργο, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Νόμιζα πως ήσασταν Γάλλος και θα σα απαντούσα έτσι αναλόγω. Μισό λεπτό να βρω τι ερωτήσει σα. Αναφερθήκατε στο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εποφελούμε από κάθε ευκαιρία να μιλάω γαλλικά, γιατί έτσι εξασκούμε. Οπότε είτε μιλώντας μαζί σας, είτε με το μερολόγιο που κρατάω. Το γράφω στα γαλλικά για να εξασκούμε στα γαλλικά. Έχω μάθει από το σχολείο, λατρεύω αυτή τη γλώσσα και μερικές φορές η ορολογία μου έρχεται πιο εύκολα στα γαλλικά στο μυαλό μου από ότι στα αγγλικά ή στα γερμανικά. Λοιπόν, έχετε απόλυτα δίκιο ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υπάρχει στενή συνεργασία. Προς το παρόν, δεν μπορώ να σας εγγυηθώ ότι αυτό θα γίνει. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω από τώρα, ως υπουργό ε, Εξωτερικών Υποθέσεων που είμαι υπεύθυνη και για την αναπτυξιακή συνεργασία και ως προεδρεύουσα, μπορώ να σας πω ότι είμαι έτοιμη να ξανάρθω εδώ και να είμαι στη διάθεσή σας για αυτό το διάλογο. Αν χρειαστεί, Μπορεί να μην είναι σαν το σημερινό, αλλά πάντως να ξέρετε ότι είμαι στη διάθεσή σας. Είτε να ξανάρθω εδώ, αν χρειαστεί, αν θέλετε, αλλά και στο γραφείο μου και οι συνεργάτες μου είναι στη διάθεσή σας. Έτσι ασκώ ε, το επαγγελμά μου και στην ε, Αυστρία. του βουλευτές στην Αυστρία του υποδέχομαι στο γραφείο μου, πηγαίνω στο κοινοβούλιο και τον θέλω αυτό το διάλογο πάρα πολύ. Μόνο έτσι δημιουργούνται νέες ιδέες. Αναφερθήκατε επίσης το στόχο του 0,7% από τον προϋπολογισμό και την αναπτυξιακή βοήθεια. Και η δικιά μου χώρα είναι μεταξύ των χωρών που δεν έχει ακόμα πετύχει αυτό το στόχο. Υπάρχει η τάση. Ξέρω ότι δεν φτάνει. Το ξέρω ότι δεν θα είναι ικανοποιητική η απάντησή μου. Αλλά ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρώσεις μας. Και όσο μέλος των Ηνωμένων Εθνών μπορώ να πω, για τη χώρα μου, ότι ξαναμπήκαμε στον ε, κατάλογο των ε, χωρών που πληρώνουν, γιατί πληρώσαμε έγκαιρα τους λογαριασμούς μας. Και παρά τις πιέσεις που υπάρχουν, τους περιορισμούς, τα προγράμματα λιτότητας κλπ. Κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι κάποιοι λογαριασμοί θα πληρωθούν όπως γινόταν μέχρι τώρα. Δεν είμαι από αυτούς που λένε «Α, κόβουμε ένα 15% από παντού». Όχι. Μπορώ να το κάνω, αλλά έχετε δίκιο με την κριτική σας. Θα προσπαθήσω ακόμα καλύτερα. Δεν λέω ότι θα πετύχουμε τον στόχο, όπως θα έπρεπε, αλλά θα παραμείνουμε σε διάλογο μεταξύ μας. Επόμενη ερώτηση ήταν της κυρίας Χόιμπου. Σας ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στο πρόγραμμα του Συμβουλίου και θα ήθελα λοιπόν να σας απαντήσω και να σας πω πως ε, φυσικά και η ε, Θέλουμε να διατηρηθεί η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Βρισκόμαστε σε διάλογο με τις ε, τρίτες χώρες. Υπάρχει ε, διάλογος, όμως ε, δεν αρκεί. χρειάζεται τότε περισσότερα. Το σύνθημα της Προεδρίας μας είναι η Ευρώπη που προστατεύει και η Ευρώπη που νοιάζεται. Η ανθρωπιστική βοήθεια, λοιπόν, για εμάς είναι μεταξύ άλλων και όχι αποκλειστικά ένα μέσο αντιμετώπιση ε, φυσικών ε, καταστροφών ή καταστροφών και άλλα σε καμία περίπτωση δεν ε, εξαρτάται από προϋποθέσεις. Το έχω πει. Στην περίπτωση του Κονγκό, της Εμένης, της Συρίας, η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είχε καμία προϋπόθεση για επανεσδοχή, προσφύγων, επιστροφές κτλ. Αυτό δεν συνέβη. Η ανθρωπιστική βοήθεια για μένα είναι βοήθεια που πρέπει να δίνεται χωρίς καμία προϋπόθεση. Αναφερθήκατε στη συμφωνία επανεισδοχής με πολλές τρίτες χώρες ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από δύο χρόνια ε, υπεγράφει μια συμφωνία τέτοια με το Αφγανιστάν. Δεν έχει εφαρμοστεί η συμφωνία αυτή έτσι όπως είχε προγραμματιστεί. Όμως συμφωνήσαμε πως τα μέσα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν θα πρέπει να εφαρμοστούν. Υπάρχει δηλαδή μία λογική αμοιβαιότητας, ε, quid pro quo. Όμως επαναλαμβάνω ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Μπορώ να πω δηλαδή πως ε, τους τελευταίους 7 μήνες ε, δεν δημιούργησα, δεν έθεσα προϋποθέσεις για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Μετά, επόμενη ερώτηση. πάνω κάτω το ίδιο θέμα, αλλά θα μιλήσω αγγλικά, ίσως είναι και πιο εύκολο για σας. Για να σας απαντήσω λοιπόν, ε, αναφερθήκατε στη σελίδα μου, στη Wikipedia αλλά να σας πω ότι σε περίπτωση μπορείτε να καταλάβετε γερμανικά θα σας ε, σύστηνα να διαβάσετε όλο το βιβλίο. Το 2012 λοιπόν έγραψα ένα βιβλίο το οποίο ήταν υποψήφιο για το, για το βραβείο καλύτερου επιστημονικού βιβλίου με γερμανικό τίτλο «Η τεστοστερόνη κάνει πολιτική, η τεστοστερόνη οδηγεί σε εξουσία». Το βιβλίο αυτό βασίζεται εξ ολοκλήρου ε, σε πηγές. Δεν είναι πολεμική, και το αναφέρατε λες και ήταν. Ε, μπορείτε νομίζω, έχετε ένα ταλέντο να παίρνετε και να διαστρεβλώνετε λόγια. Οι διερμηνείς σας ενημερώνουν ότι λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων ε, που συνεχίζονται για 37η μέρα η διερμηνία θα σταματήσει εδώ. Uh, it's fact-based.